I think we can start. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Oh. Yeah, Ja, schönen guten Καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω όλους θερμά στη συνεδρίασή μας. Μπορούμε να εκρίνουμε την ημερήσια διάταξη εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχει μια αντίρρηση από δική μου πλευράς. Διότι θα συζητήσουμε τους τριμερείς διαλόγους και κλεισμένων των θύρων, αλλά σήμερα το πρωί Ε, έμαθα ότι έχουμε ένα ε, νέο αποτέλεσμα, οπότε αμέσως μετά την ε, ψηφοφορία θα μας ενημερώσουν οι δύο εισηγητές. Μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας, της 26 Μαρτίου και Κατόπιν έχουμε την ψηφοφορία, έκθεση του Dieter Lebrecht Koch, να κάνουμε μία δοκιμή και βλέπουμε ότι το ΕΛΚ έχει πάλι ένα μέλος παραπάνω από ό,τι πρέπει. Αρχίζουμε, ξεκινάμε την δοκιμαστική ψηφοφορία να δούμε αν έχει ένα επιπλέον μέλος το ΕΛΚ. 40, 40. Also alle, die hier sind, haben abgestimmt und es ist keine über den Durst. Herzlich. Ψήφισαν όλοι οι παρόντες. Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Δεν υπάρχει κάποιο περισσευούμενο μέλος. Συμβαστική ψηφοφορία 1. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 όχι no vote, ε, τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπάρχει καμία αντίρρηση όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές, να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ, υπέρ. Μάλλον αρχίζει η ψηφοφορία, διορθώνει ο Πρόεδρος. 76, τροπολογία 76. Λήξη της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Δεν έχουμε αποχές. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 16 υπέρ, 24 κατά και 2 αποχές. Συμβαστική 10 υπέρ κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ. Εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Συμβιβαστική τροπολογία 10. Λήξη της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 8 κατά. Ήταν αρκετά σαφές το αποτέλεσμα. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 106, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 αποσύρεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ονομαστική ψηφοφορία. Abstimmung Λήξη της ψηφοφορίας. 40 υπέρ, καμία ψήφος κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή. και ευχαριστώ και την γραμματεία ε, και τους κοιόδης εισηγητές που φρόντισαν να έχουμε τόσες συμβαστικές τροπολογίες ώστε να επιταχύνουμε την ψηφοφορία. Ε, θα θέλατε να πείτε λίγα λόγια, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους. Υπέβαλαν πολύ καλές τροπολογίες ε, που Έκαναν πολύ εύκολη τη δουλειά μου να εκπονήσω συμβιβαστικέ τροπολογίε. Χαίρομαι και για την στενή συνεργασία με του σκιώδει εισηγητέ. Νομίζω ότι φαίνεται ότι είχαμε πολύ καλή συνεννόηση. Θέλω να ευχαριστήσω και του, τη Γραμματεία καθώς και την Σοφία από το ΕΛΚ. Ε, να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα δέκα χρόνια. Ε, ναι, μίλησε ο αισιόδοξο άνθρωπος ε, για την επόμενη δεκαετία. Έχουμε τώρα την έκθεση σχετικά με, τους, ε, με το χθεσινό τριμερή διάλογο. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Χθες ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε σήμερα στις 7 το πρωί. Οι εκπρόσωποι μας ε, είναι παρόντες, δεν έχουν κοιμηθεί. τους ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ, Ντομινίκ. Euh, bien, Πράγματι. Απριόρι, αυτός ο τριμερής διάλογος που συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα το πρωί θα έπρεπε να ολοκληρωθεί. Με την επιφύλαξη βέβαια ότι θα συμφωνήσουν τα κοινοβούλια, το Συμβούλιο κτλ. Για το μηχανισμό του λεγόμενου Ταμείου Juncker για να συνοψίσω τα δύο θέματα που εντάσσονται στην αρμοδιότητά μας βάσει του άρθρου 54. Η Ινές θα μας μιλήσει για τη διακυβέρνηση και εγώ θα μιλήσω για το οικονομικό σκέλος. Όπως γνωρίζετε, για το μηχανισμό εγγυήσεων ύψους 21 δισεκατομμυρίων, 16 δισεκατομμύρια θα δοθούν από το Κοινοβούλιο. Και 10 δις από τα 16 θα απελευθερωθούν, θα μπουν στο τραπέζι από το προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Και υπάρχει μία απαραίτητη ανάγκη, αυτά τα 8 ή 10 από τα 16, 8 μάλλον, να προσδιοριστούν με ακρίβεια στο κείμενο έτσι ώστε να είναι αμετάκλητη αυτή η απόφαση. Να υπάρχει δηλαδή υποχρέωση προεπιλογής των κεφαλαίων αυτών. Τώρα, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν και του Συμβουλίου, η συμφωνία ήταν δύο δις να πάρουμε από το περιθώριο ευελιξίας δηλαδή τον προϋπολογισμό του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και ότι όλα αυτά σχετίζονται με, τον, τον ορίζοντα 2020 και το Connecting Europe Facility, τη διευκόλυνση συνδέοντας για την Ευρώπη. 3,3 δις λοιπόν. Τα πήραμε από το Connecting Europe Facility και 2,7 δις τα παίρνουμε από τον ορίζοντα 2020. Έτσι έχει η κατανομή. Εξαιρετικά δύσκολες συζητήσει για το οικονομικό σκέλος, διότι όταν ξεκίνησε ο τελευταίος τριμερής διάλογος χθες το βράδυ στις 7, η θέση του Συμβουλίου δεν είχε αλλάξει. Παρέμεναν στι θέσεις τους. 6 δι από τα ταμεία επί τη ουσία και 2 δι ε, στο περιθώριο. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο αποδεκτό από εμά. Η πρόταση που βάλαμε στο τραπέζι εμεί σε συμφωνία με την Επιτροπή Προϋπολογισμού ήταν να κατανεμηθεί η προσπάθεια σε 4 δις και 4 δις. 4 δις για τα ταμεία, για τα κονδύλια μάλλον, και 4 δις για το περιθώριο. Παραμένει η θέση του Συμβουλίου για κατανομή 6-2. 6 δις και 2 δις δεν θα σας πω ότι διημήθη, αλλά τελικά η τελική πρόταση που μπορεί να γίνει αποδεκτή εάν εσείς συμφωνείτε και γι' αυτό ζητούμε συμφωνία με την επιφύλαξη, ε, με επιφύλαξη ε, στην συμφωνία που προτείνει η Κομισιόν είναι δηλαδή ότι προσπαθήσαμε να έρθουμε σε μια συμβαστική λύση 5 δις και 3 δις. Δηλαδή ανακτήσαμε ένα δις. Αυτό το δις κατανέμεται 50-50% μεταξύ του διευκόλυνση συνθέτοντας στην Ευρώπη και του ορίζοντα 2020, όμως ό,τι έχει να κάνει ε, με το Connecting Europe ε, τα 500 εκατομμύρια επανέρχονται στις μεταφορές. Άρα αυτό μας συνέφερε περισσότερο από την κατανομή 58-42 ε, ο προρατά αναλόγως δηλαδή. Και γι' αυτό προτιμήσαμε να βρούμε αυτή την συμβιβαστική λύση και έτσι αντί να ανακτήσουμε 430 εκατομμύρια θα ανακτήσουμε 500 εκατομμύρια τελικά για τις μεταφορές. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση για τη χρηματοδότηση. Υπάρχει μια προσαρτημένη πρόταση σε παράρτημα που έγινε από το Συμβούλιο. Και εκεί πάλι έχουμε, δώσαμε τη σύμφωνη γνώμη μας με επιφύλαξη. Τι λέει η πρόταση. Μέσα στο μηχανισμό ε, Connecting Europe Facility, θα το θυμάστε, υπήρχαν χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα ή ξεχωριστά με τις επιδοτήσεις από τα κράτη-μέλη. 2 δισεκατό εκατομμύρια τέτοιου ύψος, το ύψος των ε, χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων. Δεχθήκαμε λοιπόν τα 500 εκατομμύρια των χρηματοδοτικών εργαλείων να μεταφερθούν και να μεταμορφωθούν σε ενισχύσεις, σε επιδοτήσεις, grants. Μειώσαμε το μέρος των χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι παρόντα. Η Κομισιόν μπορεί να κάνει δήλωση να πει ότι δεν θα ε, εξαντλήσει το 100% των χρηματοδοτικών εργαλείων και το καθεξής μέσων. Εάν συμφωνείτε λοιπόν 5 εκατομμύρια επί ε, των, ε, των funds και 3 εκατομμύρια στο περιθώριο. σα είπα τα νούμερα για το Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη και τα 500 εκατομμύρια θα ξαναπάνε στις μεταφορές. Κατανομή προβλέπεται στο κείμενο αναλόγως με τις γραμμές που έχουν εντοπιστεί στο συνδέοντα την Ευρώπη, στη διευκόλυνση αυτή. Αυτά συνοπτικά για τον τριμερή διάλογο. Να σας πω ότι ήταν ε, κατεξοχήν ο πιο δύσκολος τριμερής διάλογος στον οποίο έχω παραστεί ποτέ μου και ε, συνεχώς η Επιτροπή ήταν στο πλάι του Συμβουλίου Δηλαδή τελικά δεν αντιμετωπίζουμε τριμερή διάλογο, αλλά διάλογο μεταξύ ημών από τη μία με ήττα και από την άλλη να είναι η Κομισιόν και το Συμβούλιο μαζί. Και αυτό πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή που θα μας μιλήσει για τη διακυβέρνηση εξίσου ακαθόδες ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην Ινέσα Γιάλα Σέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε δεδομένων των συνθήκων. Όπως είπε και ο συνάδελφος Ρίκε, δεδομένων των δυσκολιών από τις οποίες ξεκινήσαμε. Είχαμε ένα μπλόκα απέναντι στο Κοινοβούλιο, το οποίο μπλόκα παρτιζόταν από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ήταν λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο να φτάσουμε στο τέλος. Ε, πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς. Η Επίτροπος Γεωργίευα από το δημοσιονομικό σκέλος ε, θέλησε να διευρύνει το πεδίο. Είδαν ότι το Κοινοβούλιο ήταν ενωμένο και αυτό είναι, ήταν εξαιρετικά δύσκολο αλλά και εξαιρετικά θεμελιώδες. Από τότε και από τη στιγμή που είδαν ότι το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο, τότε άρχισαν τη συζήτηση για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα χωρίς να πλήξουμε τα άλλα προγράμματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα αυτού του ταμείου. Και νομίζω ότι υπάρχει τρόπος ε, να ε, μην ξεκινήσουν αυτά αργότερα, αλλά να ξεκινήσουν το 2015, κυρίως τα grants, οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις. Το Συμβούλιο αυτό το οποίο ήθελε είναι να μειώσει τα κριτήρια βάσει των οποίων το ΕΦΣΙ θα αποφασίσει για τα διάφορα μεγάλα έργα και εμείς βρήκαμε μια διατύπωση ε, through, δηλαδή να φτάσουμε μέχρι το τέλος, ενώ το Συμβούλιο ήθελε πιο πολύ particular, συγκεκριμένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς μιλούμε για το πλαίσιο, ενώ το Συμβούλιο ήθελε το in particular, το ιδιαιτέρως, για, επειδή ήθελε αυτά τα δύο μέσα να ασχολούνται με ένα πολύ μικρό πεδίο. Άρα, βρήκαμε μια ενδιάμεση συμφωνία. Μειώσαμε την αυθαιρεσία της ε, διοχέτευσης ε, των χρημάτων όπου να είναι με το in particular πιο συγκεκριμένα γίνεται εκεί λόγος π.χ. για την αστική πολιτική και από την άλλη έχουμε τα hubs που συνδέονται με το δίκτυο. Είναι ένας τρόπος διεύρυνσης mm. του δικτύου σε όλα τα θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης. Το Κοινοβούλιο θέλει να μπορεί να ελέγξει τις διαδικασίες και διατηρήθηκε ότι το ότι και πρέπει να το εξηγήσει κανείς το Συμβούλιο ότι πρέπει να έχουμε έλεγχο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγχει ετησίως το σύστημα χρηματοδότησης έπρεπε να εξηγηθεί στο Συμβούλιο το γιατί αυτού, αλλά τα καταφέραμε. Και στις διάφορες επιτροπές θα μπορεί το Κοινοβούλιο να ελέγχει και σε διάφορες πλατφόρμες, δεν θα μείνουμε σε εθνικό επίπεδο και σε εθνικές τράπεζες μόνο, αλλά θα δοθεί πρόσβαση και σε άλλους εταίρους, π.χ. περιφερειακές, τοπικές τράπεζες τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Διευρύνθηκε δηλαδή η δυνατότητα συμμετοχής. Και τέλος, ως προς το Σύμφωνο Σταθερότητας. Μεγάλος καυγάς, διότι το Συμβούλιο δεν ήθελε καν να ακούσει να γίνεται λόγος για την υποχρέωση π.χ. της Κομισιόν, όπου κατ' εξαίρεση τουλάχιστον θα πρέπει να τίθεται το θέμα της συνεισφοράς των κρατών μελών ή των εθνικών διοικήσεων για τη συμμετοχή στο ΕΦΣΥ. Ε, δεν ήθελε λοιπόν να γίνεται λόγος ότι, για το ότι αυτές οι συνεισφορές θα είναι εκτός των αυστηρών κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να ήταν με το Συμφώνο Σταθερότητας τα κριτήρια αυτά, ε, θεωρεί το Συμβούλιο. Και τελικά ε, θα υπάρξει δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό καταφέραμε, και σε ένα εκτιμώντα, σε μια αιτιολογική σκέψη θα αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει δήλωση για τη δυνατότητα εξαίρεση χρησιμοποίησης αυτών των επενδύσεων οι οποίες όταν γίνονται ε, στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ δεν θα πλήττουν τα δημόσια οικονομικά και δεν θα οξύνουν τα ελλείμματα κτλ. Ε, εκεί ε, καταλήξαμε, αυτή ήταν η συμβαστική λύση το Συμβούλιο είχε πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών και έπρεπε συνεχώς να παίρνουν τηλέφωνο οι συνομιλητές μας για να παίρνουν συνεχώς εντολές και οδηγίες για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Επομένως ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά. Ωστόσο, μπορούμε να παρουσιάσουμε και να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία γιατί θα την ελέγχουμε δημοσιονομικά ετησίως και μπορούμε και να τη διευρύνουμε για να έχουν πρόσβαση σε αυτήν οι περιφέρειες, οι πολίτες και όχι μόνο το κεντρικό κράτος και οι εθνικές ε, τράπεζες. Είναι ένας καλός τρόπος δουλειάς πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ. Βιμ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές και να τους συγχαρώ για το γεγονός ότι έχουμε συμφωνία. Περιμένω ακόμα να ακούσω τις τεχνικές λεπτομέρειες. Διότι νομίζω ότι είναι θετικό θα ήταν θετικό εάν το προσωπικό της Επιτροπής μας μπορούσε να εξετάσει τις οικονομικές συνέπειες της συμφωνίας που πετύχαμε. Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, διότι είχαμε ήδη χάσει πολλά χρήματα και οι εισηγητές έπρεπε να τα ανακτήσουν. Συγχαρητήρια και πάλι. Θα ήθελα όμως πολύ να δω τις τεχνικές λεπτομέρειες επί χάρτου, ενδεχομένως με παρατηρήσεις του προσωπικού της Επιτροπής. Και επίσης δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει το 2016. Θα μπορέσουμε να, λάβουμε πίσω όλα μας, να πάρουμε πίσω όλα μας τα χρήματα από την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη ή δεν είναι σαφές αυτό ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις των συναδέρφων Ρίκερ και Σέντερ μας δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να αγωνιζόμαστε ε, ενάντια σε ένα ενωμένο μέτωπο Επιτροπής ε, και Συμβουλίου. Ακούσαμε μία σύντομη επισκόπηση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι απομένουν κάποια ερωτήματα. Έχω να θέσω κάποιες ερωτήσεις και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο αν μπορούμε να υπερψηφίσουμε όλο το πακέτο. Αν κατάλαβα σωστά, η θέση εκκίνησης ήταν ότι θα λάβουμε 2 δισεκατομμύρια από το ε, απόθεμα και ότι έπρεπε να συμβάλλουμε με 3 ε, δισεκατομμύρια στην ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Τώρα από ό,τι κατάλαβα, 3 δισεκατομμύρια θα προέλθουν από τον ε, προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 5 θα ληφθούν τα 2,5 από το Συνέδριο στην Ευρώπη και τα άλλα 2,5 από το Horizon 2000. Ε, όχι, 2,8 και 2,2 δισεκατομμύρια αντίστοιχα, διορθώνει ο Πρόεδρος. Αυτό σημαίνει παρόλα αυτά ότι 5 δισεκατομμύρια θα λυθούν από τα ταμεία για το μέλλον, δηλαδή το συνδέοντα στην Ευρώπη και ε, το Ταμείο για την Έρευνα. Απευθύνομαι λοιπόν ε, όχι σε εσά, αλλά στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Εμείς είχαμε φανταστεί κάπω διαφορετικά τα πράγματα, δεν είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή αυτή. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, ισχύουν τα κριτήρια που έχουμε διαμορφώσει στο συνδέοντας την Ευρώπη για την έρευνα, για παράδειγμα, στα κράτη-μέλη. Και δεύτερον, τα 2,8 δισεκατομμύρια από τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη πώς θα ωφελήσουν τις μεταφορές. Διότι εγώ επιμένω ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές. Και τέλος, εάν η απάντηση στις δύο ερωτήσεις μου είναι αρνητική, τότε θα ήθελα εγώ να θέσω το ερώτημα αν θα πρέπει να υπερψηφίσουμε το πακέτο, διότι τη στιγμή που μας περιφρονούν έτσι δεν θα είναι περίεργο και εμείς να περιφρονήσουμε ε, το δικό τους αποτέλεσμα. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την εξαιρετική δουλειά τους. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι, δεν με βλέπετε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον Ντομινίκ και την Ινές για τις δύσκολες αυτές διαπραγματεύσεις. Σίγουρα δεν ήταν εύκολες οι διαπραγματεύσεις, αλλά ειλικρινά δεν περίμενα άλλο αποτέλεσμα. Έχουμε συζητήσει το θέμα επενελειμμένα στην Επιτροπή μας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι αρκετά λογικό. Έχω μια μικρή ερώτηση. Το ορίζον 2020 συζητήθηκε με την Ήτρε. Έλαβαν περισσότερη χρηματοδότηση. Μπορέσαμε σε επίπεδο κοινοβουλίου να συνεργαστούμε με την Ήτρε για να έχουμε περισσότερο συμβιβασμό και λιγότερο αγώνα για τον, τον καταμερισμό του προϋπολογισμού μεταξύ των επιτροπών. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε στο μέλλον. Θα υπάρξει μια απόφαση σε πολιτικό επίπεδο. Ως Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι θα γίνει με τα προγράμματα μεταφορών κατά την εφαρμογή του προγράμματος Juncker θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, πού θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα. Και νομίζω ότι δικό μας καθήκον είναι να κάνουμε τη δουλειά αυτή. Να εξετάσουμε δηλαδή πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Juncker στον τομέα των μεταφορών που θα ε, αντικαταστήσει την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Νομίζω ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα θέλαμε σε τακτική βάση να έχουμε συναντήσεις με τους αρμόδιους για τις μεταφορές. Πρόεδρος, να σας διορθώσω. Για το Connecting Europe θα ότι έχουμε 26 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 2,8 δισεκατομμύρια θα προέλθουν ε, από το, τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη και ε, το απόθεμα των 70 δισεκατομμυρίων είναι σχεδόν το τριπλάσιο. Ε, Πάβελ Τελίτσκα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο ήταν το έργο των συναδέλφων εισηγητών και νομίζω πως είναι σωστό να το πούμε για μένα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοήσω ε, τη στάση της Επιτροπής. Αυτό είναι ένα γεγονός. Επίσης θα πρέπει να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας, αλλά και σε άλλες Επιτροπές και αυτό στον τρόπο ήταν σχεδόν απαράδεκτος. Από αυτή τις βάσεις καταλαβαίνω πως ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση, τα αποτελέσματα ήταν πάνω κάτω αναμενόμενα. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι ο προορισμός ή η κατανομή αυτών των ε, ε, κονδυλίων ε, είναι ένα ζήτημα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ για το ΣΕΦ και το πρόγραμμα να, Juncker μιλάμε για προγράμματα μεταφορών τελείως διαφορετικής φύσης. Το γεγονός δηλαδή ότι χάνουμε από το ΣΕΦ θα πήγαινε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, άρα θα, μπορούσαμε, θα μπορούσε να περικοπεί το 10% από τα TNT, πάνω κάτω, χονδρικά. Είναι σημαντικό ποσό. Αυτό θα γίνει και θα είναι καλό να δούμε από πλευρά τη Κομισιόν συγκεκριμένη ανάλυση, λαμβάνοντα υπόψη ότι εδώ δεν πρόκειται για λογιστικά βιβλία, αλλά για λεφτά που πρέπει να ε, να τεθούν επιτάπητο, για να ακούσουμε ποια θα είναι οι εξηγήσει. Εδώ ε, λοιπόν ε, επενώ τους συναδέλφους για τη σκλήρια τους δουλειά, αλλά θα ήθελα όλα αυτά να τα δούμε και γραπτός και ίσως έτσι να μπορέσουμε να το σχολιάσουμε, γιατί είναι δύσκολο να διαβάζει κανείς νούμερα χωρίς να γνωρίζει τι έχει γίνει το μεταξύ και νομίζω πως ε, τα όσα έχουν γίνει το μεταξύ θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη δυσκολία και ίσως το γεγονός ότι να μην υπήρχε άλλη επιλογή. Πάντως σίγουρα δεν είναι τώρα σαφές Βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λεπτομερώς με τον Ντομινίκ. Να δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες, να τις αναλύσουμε και να το ξανασυζητήσουμε για να καταλήξουμε σε μια θέση. Σας ευχαριστώ. Kerrankin voisin melkein sanoa, arvoisa puheenjohtaja, että olen lähes sanaton. Εγώ θα ήθελα να πω ότι κάποιες φορές μένω άφωνη. Γιατί η ομάδα μας αυτές τις διαπραγματεύσει πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε. Και από την άλλη πλευρά είναι καλό το γεγονό ότι ούτως ή άλλως οι μεταφορές φέρνουν περισσότερα χρήματα από οτιδήποτε άλλο στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή μας και να τους, ευχαριστή και να, τους εισηγητές μας και να τους ευχαριστήσουμε για το τι κατάφεραν. Ελπίζω ότι οι μεταφορές θα εξακολουθήσουν να συγκεντρώνουν ε, κονδύλια για τις νέες καινοτομίες και για τα πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα που κυκλοφορούν. Πρέπει να συνεχίσουμε όπως και παλαιότερα Και θα πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά το τι γίνεται για να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Δεν ξέρω ακριβώ τώρα πώς να το πω. Πάντως, δεν ξέρω αν έχουμε ότι κάτι να κερδίσουμε ε, αυτή τη φορά. Πάντως, αν υπήρχε κάτι, σίγουρα το έχετε καταφέρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Καρή Μαντελή. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους ηγητές ε, γιατί έχουν κεντήσει. Ε, πρέπει δηλαδή να διαπραγματευτεί λέξη τη λέξη και νούμερο τον αριθμό τον αριθμό. Μπράβο σας λοιπόν. Όμως το σχέδιο Juncker είναι κομμάτι της καλύτερης νομοθεσίας του Better Legislation είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε στο μέλλον με τις καλύτερες πρακτικές. Κατά τη γνώμη σας, ως εισηγήτω, Ίσως για το... Πραγματικά πιστεύετε ότι αυτό εντάσσεται στην καλύτερη νομοθεσία. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως ε, πόρο απέχει. Αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας. Γιατί ακριβώ έτσι παρουσιάστηκε. Λες και είναι η καλή πρακτική. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον όλοι. Έπειτα, μπορείτε εσείς να με καθισχάσετε, κύριε ε, ότι στο άρθρο 5.2 θα μείνει που λέει και αναφέρει ακριβώς όλα τα οριζόντια προγράμματα. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι λίγο σε αυτό το σχέδιο Juncker έχουμε αυτή τη, ε, τη γραμμούλα. Εγώ θαυμάζω την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αλλά την έχουμε. Και σε αυτό το κομμάτι μεταφορές έχουμε ό,τι χρειάζεται για τις κλιματικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ και πάλι μπράβο σας. Ευχαριστώ, Πέτερ Λόντγκρεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την νυχτερινή δουλειά σας. Ελπίζω να κοιμηθείτε καλά μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης ε, για να αντισταθμίσετε την έλλειψη ύπνου. Δεν ε, έχω αντίρρηση όσον αφορά τις ε, την εξοικονόμηση και επίσης ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, δυστυχώς τώρα δεν μιλάμε για εξοικονόμηση, μιλάμε για ανακατανομή. Θα περιμένω όμως να δω τις πρακτικές λεπτομέρειες ε, σε γραπτή μορφή για να έχω μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαρίν ask, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ο Ντομινίκ να μας πει δύο λόγια για την προσθήκη στο άρθρο 8. Είναι σημαντικό η χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ να αποφασιστεί κατά την ε, ε, τακτική ετήσια διαδικασία εξέτασης του προϋπολογισμού. Μπορούμε να ε, απελευθερώνουμε κονδύλια για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και για τον ορίζοντα 2020 και να το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο. Υπάρχει προσθήκη σχετική στο άρθρο 8, παρακαλώ να τη σχολιάσετε και με βάση, αυτόν μπορούμε να, με βάση αυτά μπορούμε να δεχθούμε και να συμφωνήσουμε ε, με αυτό που μας προτείνεται, που δύσκολα επιτεύχει. Dziękuję bardzo, przewodniczący. Rzeczywiście... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συζητητές και για τη σκληρή νυχτερινή δουλειά που κάνανε. Επί της ουσίας, νομίζω ότι εδώ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου αναζητείται απεγνωσμένα ένας δρόμος για να χρηματοδοτηθεί μια ιδέα του Ιούνκερ που θα πρέπει να δώσει περισσότερη ορμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά όμως μεταφέρουμε πόρους ε, από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και τους πόρους ε, της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Το θέμα όμως είναι και η γεωγραφική κατανομή πού θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα και η κατανομή θα γίνει αναλογικά ή επιλεκτικά. Και επίσης έχουμε και μία τομεακή κατανομή. Θα πάρουμε χρήματα από όλους τους τομείς ή θα επικεντρωθούμε σε κάποιους τομείς μόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το γενικό μας όραμα, καθώς και όσον αφορά την αξιολόγηση των ε, συμφορήσεων και τα αποτελέσματα που περιμένουμε από την επένδυση των πόρων αυτών. Θα πρέπει σύντομα να είναι σαφές ποια προγράμματα θα τροποποιηθούν ή ποια θα παθούν. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Θέλουμε να δώσουμε ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε όμως να έχουμε το δικαίωμα να συζητήσουμε τις συνέπειες αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μας Μιλάνο Σαλίνη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει και συμφωνώ με πολλά από τα όσα άκουσα και τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν. Ένα στοιχείο, ένα επίκαιρο δηλαδή στοιχείο, λέει ότι η πρώτη Ιταλική επένδυση που έχει ενταχθεί στο σχέδιο Juncker είναι μια σημαντική επένδυση βιομηχανικού τύπου. Στην βιομηχανία, στη Χαλιβουργία μάλιστα και μάλιστα στην επαρχία μου, την επαρχία της Κρεμόνα, στη Λομβαρδία. Ήδη λέει υπογράφηκε και ήδη την υπέγραψε η, Μπέη, η ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με συγχωρείτε. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην Ιταλία, όπου λεγόταν ότι πιθανότατο μέγα τμήμα του σχεδίου Juncker θα αφιερωθεί στη βιομηχανική ανάπτυξη και πολύ λίγα θα δοθούν στις μεταφορές, γιατί οι μεταφορές δεν αποδίδουν ε, γρήγορα σε σχέση με το κεφάλαιο που επενδύεται. Εμένα δεν με πειράζει. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Βιομηχανία. Αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η βιομηχανία θα πρέπει με άλλο τρόπο να αναζωογονηθεί. Τα δημόσια κονδύλια θα πρέπει να κατευθυνθούν στα δίκτυα. Είτε είναι TEN-T, TEN-E ή TEN, όπω θέλετε πείτε τα, πάντω πρέπει να πάνε στα δίκτυα χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε σημεία επαφής με το εκτός της Ευρώπης, δηλαδή λιμάνια και αεροδρόμια, τεράστιο δυναμικό ανάπτυξη στην Ανατολική Ευρώπη που αυτή τη στιγμή δεν συνδέεται επαρκώς με την Κεντρική Ευρώπη. Αυτά όλα λοιπόν όπως είπαν οι συνάδελφοι και πολλοί εισηγητές πάνε στην κατεύθυνση του να στηρίξουν τελικά με λάθος μέσα κάτι το σωστό. Πρέπει λοιπόν να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ Ρώσο Νταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη δουλειά που έκαναν, όμως δεν θεωρώ πως είναι νίκη μας. Γιατί Εδώ η γνώμη του Κοινοβουλίου και η γνώμη ε, θεωρείται μηδενική. Την αγνοούν τελείω. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο ακολουθούν το δρόμο του. Εμεί θα πρέπει να ικανοποιηθούμε με το να σώσουμε ένα δι από τι επενδύσει του ΕΦΣΥ. Είναι ε, κάτι ελάχιστο. Καλύτερο από το τίποτα, αλλά όπω ήδη είπαν οι συνάδελφοι και, και ο μόλι προηγούμενο από μένα συνάδελφο, ε, ε, υπάρχουν ήδη, η, η, η Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων έχει ήδη τα προγράμματα και χειρίζεται εγκρίνη. Εμεί δεν έχουμε ακόμα βγάλει τη δική μα ονομοδότηση και εκείνοι ήδη ξέρουν τι θα χρηματοδοτήσουν. Ε, ποια σχέδια και μάλιστα τη χαλιβουργία για παράδειγμα. Μα αυτό γίνεται και στην Ιταλία, αλλά σίγουρα θα γίνει και για άλλες χώρες. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η γνώμη μας ε, ε, τελείως αγνοείται. Λάθος κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τους εισηγητές. Πιστεύω ότι σπάνια έχουμε ακούσει τόσο θετικές παρατηρήσεις, ακόμα και αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι εισηγητές κατάφεραν ε, το, μέγιστο, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ε, τους ευχαριστώ και τους ευχαριστώ που παρέμειναν ε, εδώ στο Κοινοβούλιο παρότι τελείωσαν στις 7 η ώρα το πρωί για να έρθουν να μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Το αποτέλεσμα του, του ημερούς διαλόγου θα διανεμηθεί σε όλους ώστε να είναι σαφή και τα νούμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι πρόκειτο για τριμερή διάλογο. Επρόκειτο για μονομαχία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο από τη μία και το Συμβούλιο και, το και την Κομισιόν από την άλλη. Και μου φαίνεται ε, λίγο περίεργο αυτό, διότι το Συμβούλιο δεν ε, δίνει καθόλου ε, χρήματα για αυτό το πρόγραμμα των 350 ε, δισεκατομμύριων. και η Κομισιόν πήρε το μέρος του Συμβουλίου. Αυτό είναι κάπως περίεργο. αλλά έχουμε εδώ εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Ε, Μήπω ε, θέλετε να πείτε λίγα λόγια, παρακαλώ. Με πιάσατε λίγο εξαπίνης, κύριε Πρόεδρε, γιατί ανακαλύπτω, όπως και εσείς, τώρα τις λεπτομέρειε της έκβασης του τριμερούς διαλόγου. Να πω δύο λόγια ωστόσο. Πρώτον, το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ανέκαθαν ήμασταν υπέρ της στήριξης αυτού του ταμείου και της σημασία του. Και πρέπει να κοιτάζουμε και πέρα από τις μεταφορές και να έχουμε υπόψη μας το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνειδητοποιούμε πόσο καθοριστική σημασία, πόσο αποφασιστική είναι αυτή η απόφαση τελικά. Για χρόνια αγωνιζόμαστε με τα κράτη-μέλη και με το Συμβούλιο για να έχουμε ένα αφιερωμένο μέσο ειδικό για να χρησιμοποιηθεί για τις επενδύσεις σε υποδομές και σε άλλα μεγάλα έργα με ορίζοντα το μέλλον. Δεν έχουμε ένα τέλειο ταμείο, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα στέρεο μέσο, ένα στέρεο εργαλείο. Και Πιστεύω ότι η δουλειά σας συνέβαλε, ο εισηγητής συνέβαλε εξαιρετικά. Όλα τα συστατικά λοιπόν υπάρχουν και μπορούμε να έχουμε συμφωνία, μπορούμε να βελτιώσουμε την αρχική πρόταση και όλα αυτά αναπτύχθηκαν μέσα ε, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή εγώ περιμένω καλύτερα κριτήρια επιλεξιμότητας. Δεύτερον, καλύτερος ορισμός του τι σημαίνει πραγματικά το additionality, προσθετικότητα αν θέλετε, και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων να αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια για έργα υψηλότερου ρίσκου, όχι παραδοσιακά, και αυτό είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτο αν συμβαίνει και από τη δημοσιονομική σκοπιά ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Ε, να φέρετε ένα εκατομμύριο ευρώ, λέει ο μιλητής, ε, για grants, για ενισχύσεις, να, να το πάτε εκεί, μάλλον ένα δις εννοεί. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά και καλά ε, έργα, επομένως αυτό το έξτρα ένα εκατομμύριο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος και θα αξιοποιηθεί πολύ σωστά, λέει πάντοτε ο μιλητής. Τέλος, αναλύοντας τη δυνατότητα της υφιστάμενης ε, διαδικασίας του προϋπολογισμού ε, πρέπει να δούμε αν όλα αυτά συνάδουν, είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι ε, όταν θα έρθει το σημείο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό θα είναι εξαιρετικά θετικό. Προτεραιότητά μας τώρα είναι να είμαστε σίγουροι ότι θα αξιοποιήσουμε αυτό το ταμείο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα ήθελα με τη δική σας επιτροπή να περάσουμε λίγο χρόνο για να σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πώς έχει ε, εξετάσει όλα τα έργα τους διαδρόμους των διευρωπαϊκών δικτύων 10T Corridors να δούμε ποια είδους έργα θα είναι επιλέξιμα για αυτό το ταμείο και ε, να προσπαθήσουμε να έχουμε μία πρώτη λίστα, αν θέλετε, των πιο χρήσιμων έργων ε, που είναι χρήσιμα για το κόσμο των μεταφορών. Γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι οι υποδομές στις μεταφορές μπορούν να επιδοτούνται μόνο με τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά απλουστευτικό και εύκολο. Μπορούν να τύχουν και άλλες χρηματοδότησες. Ευχαριστώ. Κύριοι συγητές, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Θα ήθελα να απαντήσω, λέει ο κύριος Ρικέ, ε, στις ερωτήσεις επί της ουσίας και στη συνέχεια οι νέες για τα θέματα διαφάνειας, ορατότητας και τα λοιπά, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πράγματι λοιπόν, ε, σημειώνω ότι είναι πολλές οι αντιδράσεις από πλευρά συναδέλφων. Πολλοί θέλουν να πάρουν το λόγο και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Δείχνει το πνεύμα που μας διέπει, δείχνει το πόσο δύσκολη είναι η συζήτηση ούτως ή άλλως. Τώρα, για να απαντήσω στα δημοσιονομικά ερωτήματα που μου τέθηκαν, τα θέματα του προϋπολογισμού, κάτι το πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι το εξή. Στην αρχή η πρόταση προέβλεπε δύο δις από τα περιθώρια, από το περιθώριο και παρουσιάστηκε από το Συμβούλιο ως, ως η δική του συμβιβαστική πρόταση. Δηλαδή δεν παρουσιαστήκε ως σημείο κίνησης αλλά ως συμβιβαστική πρόταση μαζί με την Κομισιόν. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι και φυσικά δεν μας αρέσει το Συμβούλιο θεωρεί ότι τα περιθώρια ίσουνται με χρήματα. Κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό. Και όταν συζητούμε για να πάρουμε άλλο ένα δις από τα περιθώρια το Συμβούλιο θεωρεί ότι παίρνουμε ένα δις από τη δική του τσέπη. Και αυτό είναι ε, μεγάλη δυσκολία. Και μάλιστα, από πίσω υπάρχουν οι απότερες ε, δημοσιονομικές συζητήσεις. Ό,τι δηλαδή στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Και ε, περάσαμε ώρες προσπαθώντας να ορίσουμε ποια είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση. Και είπαμε λοιπόν τελικά θα κάνουμε 5-3, 5 δις από το ταμείο, 3 δις από το περιθώριο. Όμως η άσκηση του προϋπολογισμού είναι ετήσια, δηλαδή η χρήση οικονομική είναι ετήσια στον προϋπολογισμό. Άρα πρέπει να έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες και να πούμε δεν θα ξεπεράσουμε τα 5 δις π.χ. στο σύνολο των κονδυλίων των διαθεσίμων αλλά στις αιτήσει κατανομές, στην διάμεση αναθεώρηση δύο είναι οι δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε ή θα κινητοποιήσουμε περισσότερο τα περιθώρια και άρα ε, κατά αντίστοιχο ποσό θα μειώσουμε την προσφυγή στα κονδύλια, στο funds το 2 δις και 8 δις είναι το μέγιστο. Μπορούμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε περισσότερο τα περιθώρια ευελιξίας, πρώτον, και δεύτερον, ενδιάμεση αναθεώρηση σε μια στιγμή κατά την οποία πράγματι μπορεί να ξανανοίξουν και άλλα κεφάλαια ε, δημοσιονομικά ή του προϋπολογισμού αν θέλετε. Άρα, το Συμβούλιο θεωρεί ότι μας πήρε δύο δις και καλός, αλλά έχουμε όμως δυνατότητα reflow να επανέλθουμε στα περιθώρια. Εάν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, παρόλο που είναι αυτό περίπλοκο. Να απαντήσω στο τι βάλαμε τελικά στο κεφάλαιο 8. Θα σας διαβάσω τις τέσσερις αυτές σειρές, τις τέσσερις γραμμές εξαιρετικά σημαντικές κατά τη γνώμη μου τα ετήσια κεφάλαια από το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραχή αυτού του Ταμείου Εγγυήσεων θα εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονισμό 3011 το 2013, εάν δεν έκανε λάθος τη διερμηνία σας, και ε, λαμβάνοντας υπόψη το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-2020. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό στο κείμενο να πούμε ότι είναι μια ετήσια υλοποίηση του προϋπολογισμού και θα τη χάνει αναθεώρηση, revision. Και περάσαμε ώρες να σας πω στο να συζητάμε τη διαφορά μεταξύ του revision και του review. Ε, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι τα, είναι χαμένα τα πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ένα δις που πήραμε, που αποκτήσαμε, πέτε το όπως θέλετε, μετά τον τριμερή διάλογο. 500 εκατομμύρια από τα περιθώρια ευελιξίας του 2014 που δεν αξιοποιήθηκαν. Το Συμβούλιο όμως είπε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, δέχθηκε να χρησιμοποιήσει 500 εκατομμύρια από το περιθώριο ευελιξίας για το 2015. Το περιθώριο ευελιξίας του προϋπολογισμού του 2015 αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 1 δις 600 εκατομμύρια. Αλλά τελικά το περιθώριο που θα μείνει θα ξεπεράσει λίγο το 1 δις κατά τη. Όμως το Συμβούλιο θέλει τα 500 εκατομμύρια. Γιατί, γιατί θέλει να μειώσει ε, τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των πληρωμών και των δεσμεύσεων. Γιατί ξέρετε κάθε χρόνο κλείνει χρονιά με διάφορα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια καθυστερούμενων ή ληξεπρόθεσμων οφειλών. Πράγματα δηλαδή που δεν έχουμε πληρώσει. Θα υπάρχει λοιπόν ετήσια εκτέλεση του προϋπολογισμού με την υποχρέωση αναθεώρησης ενδιάμεσης midterm review και εκεί το Κοινοβούλιο έχει να δώσει μεγάλη μάχη και να αξιοποιήσει το θέμα της ευελιξίας. Στη θεωρία, εάν το περιοριστούμε στο άρθρο 14, θα πρέπει να έχουμε και να βρούμε κιόλας και λογικά θα συμβεί αυτό, περιθώρια από τα δικά μας ταμεία και τα δικά μας κονδύλια. Έχουμε την ελπίδα δηλαδή κάτι ακόμα να κερδίσουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα πολύ σημαντικά και θα μας τα πει η ΝΕΣ. Πώς κατανέμουμε αυτά τα ποσά στο Connecting Europe Facility. Βεβαίω, προφανώς ε, η διευκόλυνση αυτή ανοίγει δυνατότητες για τις μεταφορές και τα θέματα που μας είναι πολύ προσφυλή. Η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τις μεταφορές μέσω αυτού του πλάνου θα πρέπει να την εγκαταλείψουμε. Μπορούμε να τη στηρίξουμε, αλλά βέβαια ο όγκος του μηχανισμού είναι πιο σημαντικός. Υπάρχει, και η Νέσα σας το πει, είδαμε μετά πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις ε, τομεακές κατανομές ή τις θεματικές κατανομές. Εκεί όπου υπάρχει υπερσυγκέντρωση, μάλλον για να αποφύγουμε την υπερσυγκέντρωση τη γεωγραφική, τη αλλά σα θυμίζω ότι στις πρώτες δεσμεύσει που ανελήφθησαν ε, μάλιστα εξάντε από την ε, ΕΤΕΠ υπάρχουν ε, δυνατότητες χρηματοδότηση των μεταφορών. Δεν είναι μόνο βιομηχανία δηλαδή τα προγράμματα. Δεν θέλω να πω τώρα τα όσα θα σας πει η Ινές. Euh, Για την ερώτηση του Ισμαέλ. αν θα ξαναδούμε τα 2,8 δις που κατά κάποιο τρόπο δώσαμε στον μηχανισμό Juncker μέσω αυτού του μηχανισμού, ε, ειλικρινά δεν μπορώ να πω τι ακριβώς θα μπει εκεί, πάντως εφόσον Αν δεν καταφέρουμε να έχουμε πάνω από το 1% δεν θα τα έχουμε καταφέρει υπέροχα. Ελπίζω πολύ περισσότερο θα πάρουμε πίσω. Γιατί θα πρέπει να δεχτούμε ότι αν δεν πάρουμε τα λεφτά μας πίσω σημαίνει ότι θα έχουμε χρησιμοποιήσει λιγότερο από το 1% του μηχανισμού. Γύρω στο 30% ε, θα πρέπει να δοθεί σε υποδομές για τις μεταφορές. Ίσως όχι αποκλειστικά στο core network, ε, αυτό είναι σαφές, ε, ίσως αποκλει... όχι αποκλειστικά για τα δικά, με βάση τα δικά μας κριτήρια επιλεξιμότητα και η Νέα σας είπε και για να πω και στην Καρίμα και για τους κόμβους και για τα θέματα τα περιβαλλοντικά ε, και θα πρέπει να ξαναπάρουμε τα λεφτά μας πίσω γιατί διαφορετικά θα είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα. Αναφορές, αναφορές, ναι, ναι. Ναι, ναι, θα συντομεύσω. Είναι πολλά. Ναι, είναι αλήθεια, έχουμε και άλλα να κάνουμε. Θα το, θα το δείτε, είναι στο κείμενο και εδώ σταματάω γιατί ο, ο πρόεδρος με κοιτάει άγρια. Je Σας επιτρέπω όμως να είστε κουρασμένος. Ε, η Νέσα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο λέει ο συνάδελφος κύριος Ρικέ. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση έχουμε ενισχύσει το ρόλο του Κοινοβουλίου και την ε, φόρμουλα του προϋπολογισμού για να ξανατροφοδοτήσουμε αυτό το οποίο εγκαταλείπουμε. Δηλαδή δεν βάζουμε στο τραπέζι χρήματα cash σε ρευστέο, αλλά την εγγύηση ότι αν υπάρξουν απώλειες από το μηχανισμό θα υπάρξουν χρήματα που θα έρθουν από τη χύψη πηγή, εάν αυτό αποδειχθεί αναγκαίο. Άρα θα μπορούμε να ανακτήσουμε από τα περιθώρια μέρος αυτό που θα έχουμε ενδεχομένω απολέσει. Για φέτος ας πούμε δεν θα χρειαστεί. Γιατί με το ένα δις και με τις εγγύήσει καταφέραμε να αποφύγουμε τέτοιο θέμα. Ενισχύθηκε λοιπόν η συμμετοχή και η σημασία της συμμετοχής των μεταφορών σε όλο το μηχανισμό και ενισχύθηκε η ικανότητα του Κοινοβουλίου να ελέγχει τον προϋπολογισμό και την εκάστοτε οικονομική χρήση. Η αιτήσια γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών για τον προϋπολογισμό θα περιλαμβάνει απαραίτητο έλεγχο πιο σημαντικό από ό,τι έχουμε συνήθως διότι συνήθω εκδίδουμε γνωμοδοτήσει που υποβάλλουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών και μετά αυτή την κάνουν ό,τι θέλουν την γνωμοδότησή μας, ενώ τώρα η δική μας γνώμη θα αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ. Να πω επίση ότι σε σχέση με τα διδάγματα που αντλήσαμε, είχαμε ένα εσωτερικό καυγά με τον ορίζοντα 2020, γιατί αυτό είναι ο πιο όμορφος και δεν είναι πολύ κομψό που το λέω, αλλά με το λόμπι όλων αυτών που έχουν πάρει Νόμπελ και που θέλουν τον ορίζοντα 2020, ε, έπρεπε να αντιπαραταχθούμε και να βρούμε ένα κοινά αποδεκτό, μια κοινός αποδεκτή περίμετρο και ε, οι επιστροφές θα πρέπει να γίνουν στο σύνολο της διευκόλυνσης ε, συνδέοντας την Ευρώπη και να διατηρηθούν οι προτεραιότητες. Υπάρχει ένα βαθμολόγιο για την ε, ε, γεωγραφική κατανομή στις περιφέρειες. Πού πάνε τα κονδύλια μέσα στο έφσι και με βάση ποιες αρχές, την αηφορία, τις κοινωνικές αρχές και το καθεξής. Και τέλος, να σας πω ότι στο 5-2 με αυτό το τέχνασμα, το λεκτικό του in particular και του through διατηρήσαμε τις προτεραιότητές μας. Δηλαδή το θέμα της αστι... αστικής κινητικότητας. Κάτι το οποίο συνάδει πλήρως με αυτό που θέλει ο κύριος Γιούνκερ ο οποίος μας είπε εξ, ορχής, ότι έχει εντολή να ενισχύσει όλες τις πτυχές της αστικής πολιτικής μεταφορών. Και βέβαια, ως προς τα χρήματα που θα βγάλει από το Ταμείο της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το πιο σημαντικό είναι το θέμα της βιομηχανικής ανάπτυξης. Έχουμε την τάση να θυματοποιούμαστε και να λέμε μας τα πήραν όλα, μας τα παίρνουν και το καθεξής. Όχι, μπορέσαμε να διατηρήσουμε πολλά. Και άλλωστε η βιομηχανική ανάπτυξη δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και άρα δημιουργεί ανάγκη κινητικότητας. Γιατί τα ε, προϊόντα, για παράδειγμα, οι πρώτε ύλε που χρησιμοποιούν δεν τι ε, παράγουν στην περιοχή που βρίσκεται το εργοστάσιο, πρέπει να τι μεταφέρουν. Και άρα αυτό μα ενδιαφέρει εμά ε, ω Επιτροπή Μεταφορά. Δηλαδή, συνολικά έχουμε καταφέρει μια καλή συμφωνία. Τους βγάλαμε από την τσέπη τους ένα δις. Τους πήραμε ένα δις από την τσέπη, από την τσέπη τους Συμβουλίου. Και στις 7 το βράδυ ήταν 0 το δις που βγάλαμε από την τσέπη του Συμβουλίου. Ξεκίνησαν με τα 143 και τελικά ε, εκατομμύρια και με τελικά εμείς το ανεβάσαμε μέχρι το ένα δις είναι νίκη του Κοινοβουλίου ότι αντί για το 6-2 πήγαμε στο 5-3. Υπάρχουν ε, περιθώρια που θα αφαιρεθούν σε ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή είναι η πραγματική νίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την καταφέραμε γιατί ήμασταν ξεροκέφαλοι και δεν υποχωρήσαμε ως Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι τους δύο εισηγητές και για αυτές τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό που παρεμβάλαμε το θέμα αυτό για να ενημερωθούν όλοι. Προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Θα πρέπει να προσέξουμε το χρόνο, να επιταχύνουμε λίγο. Δίνω το λόγο στον Βίν Φαμτεκάμπ για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ ομαλή η μετάβαση από το EFSI στην Λευκή Βίβλο για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Για να εφαρμόσουμε τις ιδέες στην Λευκή Βίβλο, σίγουρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του EFSI, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέρφους για τις πολλές τροπολογίες που υπέβαλαν. Δυστυχώ, όμως ε, δεν ακολούθησαν την έκκλησή μου να μην στείλετε υπερβολικά πολλές τροπολογίες. Μου είπε όμως ο κύριος Ρικέ, μη φροντίζεις, είναι φυσιολογικός αυτός ο αριθμός τροπολογιών για μια λευκή βίβλο. 625 τροπολογίες έχεις και θα πρέπει να τις σε ένα λογικό αριθμό συμβιβαστικών τροπολογιών. Αυτό κάνουμε λοιπόν τώρα. Είχαμε ε, μία συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε άλλη μία. Και σήμερα το πρωί 7 παρα 4 πήρα μήνυμα από τον συνάδελφό μου Μπάς Έικχοτ που είπε ότι είχε περάσει όλη νύχτα συζητώντας το θέμα αυτό και γι' αυτό δεν θα ήταν σε θέση σήμερα το πρωί να συζητήσει το θέμα. Υποβλήθηκαν πολλές τροπολογίες για τη βιωσιμότητα και την οικολογική διάσταση, το πρασίνισμα των μεταφορών. Στις συμβαστικές τροπολογίες ε, έχουμε αναφέρει και τους στόχους της ε, συμφωνίας με το Συμβούλιο πέρσι. Θα θυμάστε ότι υπερψήφισαν το πακέτο για το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου και σήμερα έχει ενσωματωθεί στις συμβαστικές μας τροπολογίες. Τρίτον, ε, στις τροπολογίες δεν δίνεται πολύ βάρος το οικονομικό κέρδος ε, των μεταφορών. Ε, αναφερόμαστε περισσότερο στην δαπάνη χρημάτων ε, και όχι τόσο πολύ στο πώς μπορούμε να εισπράξουμε χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να εισπράξει κανείς τα χρήματα και μετά να τα ξοδέψει. Μπορεί άλλα πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου μας να το βλέπουν διαφορετικά, αλλά εγώ θα διαφωνήσω. Ελπίζω όμως ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να λυθούν στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Όσον αφορά την πολυτροπικότητα, ε, συμφωνούμε και αυτό εκφράζεται και στις τροπολογίες μας. Επίσης, μάλλον συγγνώμη, μπερδεύτηκα λέει ο μιλητής. Αναφερόμαστε και στην ε, μεταφορά επενδύσεων από τους σιδηροδρόμους ε, στις ε, εσωτερικές πλωτές οδούς. Το να διπλασιάσουμε τις δημόσιες μεταφορές στις πόλεις είναι κάτι το οποίο θα υποστηρίξουν πολύ νομίζω. Συνδέεται με τις εκπομπές σωματιδίων. Υπάρχει όμως εδώ το πρόβλημα της επικουρικότητας. Έχουμε όμως πόρους για την έρευνα και θα μπορέσουμε έτσι να προκαλέσουμε αλλαγές και να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. με τόσες τροπολογίες όμως δυσκολεύομαι και νομίζω ότι αρκετές από αυτές είναι θέμα επικουρικότητας. Σε όλες τις πόλεις μας υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν το ποδήλατο. Θα το δείτε αυτό και στην έκθεση της κυρίας Ντελή. Να μην ε, βλέπουμε όμως υπερβολικά ρομαντικά τις μεταφορές στις πόλεις. Πάντα θα υπάρχουν αυτοκίνητα, θα πρέπει απλά να φροντίσουμε να περιορίσουμε τον αριθμό τους. Επίσης, ε, πολλές τροπολογίες επικεντρώνονται στα κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με τις μεταφορές. Θα πρέπει να περιμένουμε εδώ τη διαπραγμάτευση άλλων πακέτων. Δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα τα θέματα στις τροπολογίες μας. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα κεντρικά θέματα της έκθεσης. Επίσης, ε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Η Ευρώπη είναι ευφυής και μπορεί να αναπτύξει σύγχρονα συστήματα, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο και μπορεί να αυξήσει την απασχόληση όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών αλλά και αλλού. Ένα παράδειγμα των κοινωνικών μέτρων έχει να κάνει με τους χώρους στάθμευσης. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό θα αποτελέσει καλό τρόπο επένδυσης των χρημάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Κλείνοντας, όπως είπα και νωρίτερα, να πω ότι είναι πολύ αναλυτικές κάποιες τροπολογίες και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις χειριστούμε. Η Λευκή Βίβλος έχει ειδικό της χαρακτήρα. Δεν είναι το ίδιο με μια αναλυτική έκθεση ή έναν αναλυτικό κανονισμό ή μια οδηγία. Θα ήθελα λοιπόν να διατηρήσω αυτόν τον χαρακτήρα της έκθεσης αυτής. Οι σκιώδεις εισηγητές είναι διατεθειμένοι να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Έχει προγραμματιστεί η ένα αναλυτικο κανονισμο η μια οδηγια θα ηθελα λοιπον να διατηρησω αυτον τον χαρακτηρα της εκθεσης αυτης οι σκιωδεις εισηγητες ειναι διατεθειμενοι να συζητησουμε τις συμβαστικες τροπολογιες εχει προγραμματιστει η ψηφοφορια για την συνεδρίαση της Επιτροπής μας του Ιουλίου, το πρωί της 14ης Ιουλίου, εάν το κάνω λάθος. Βέβαια, ε, αυτή η ημερομηνία ε, θα έρθει πολύ σύντομα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητές. Κλάουτια Ταπαντέλ, παρακαλώ. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Βήμα και τους συναδέλφους που εργάστηκαν για την έκθεση αυτή που αφορά την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα, στις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι και σίγουρα Βήμα δεν θα τα βρει εύκολα για να φτιάξει συμβιβαστικέ τροπολογίες. Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες, αλλά ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε. Γενικό σχόλιο ε, να πω ότι όσον αφορά την ποιότητα ε, των προτάσεών σας ε, έχουμε εδώ καλή ποιότητα και ελπίζω πως οι περισσότεροι συνάδελφοι θα βρουν τις ιδέες τους να αντικατοπτρίζονται στις συμβιβαστικές. Ε, χρειαζόμαστε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο θα είναι οργανωμένο γύρω από τον επιβάτη και από τη χρήση των υπηρεσιών επιβατών και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Καλωσορίζω τώρα την ιδέα για συμπερίληψη μιας κοινωνικής διάστασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο και η ομάδα μου το επιθυμούσε αυτό πολύ. Ε, οι συνθήκε εργασία και η ισότητα στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε καταθέσει τέτοιε τροπολογίε. Υπάρχουν δε κάποιε πτυχέ τι οποίε θα ήθελα να επιμείνω. Ιδιαίτερα η επιθυμία για επίτευξη συμβιβαστική που όμω δεν θα αμβλύνει τι ε, τροπολογίε που έχουν κατατεθεί να δεχτούμε και αυτή την πρόταση να, να διατηρηθεί η πρόταση για τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στην τροπολογία 66. Στο τελικό κείμενο Υπάρχουν και οι τροπολογίες που εμείς συντάξαμε για να ευθυγραμμίσουμε τους στόχους της Λευκής Βίβλου με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από τον Οκτώβριο του 2014 καθώς και με τους στόχους που έχουμε για ε, τον τομέα ETS. Ε Τώρα, για τις υποδομές και τις φυσικές υποδομές όταν μιλάμε για διατροπικότητα και για αλλαγή στους ε, τρόπους μεταφορών. Θα θέλαμε να διατηρηθεί αναφορά στην διατροπικότητα, στη χρήση δηλαδή διαφόρων μορφών μεταφορών ε, χρησιμοποιώντας το πιο, τους πιο αποδοτικούς ως προς την ενέργεια ε, τρόπους μεταφορών. Ελπίζω πως αυτό δεν θα ξεχαστεί και για την παράγραφο 6 θεωρούμε ότι στις συμβιβαστικές θα πρέπει να μείνουν τα κείμενα των τροπολογιών που επιμένουν για τη δημιουργία αδιάκοπων μεταφορών για τους επιβάτες. Ε, θα θέλαμε να συντάξουμε λοιπόν συμβιβαστικές που θα καλύπτουν όλες τις στοιχείες που συζητήθηκαν σήμερα το πρωί και αυτές οι συμβιβαστικέ δεν θα πρέπει να καταργήσουν τις αναφορές στο Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο Μεταφορών και στα προγράμματα βιώσιμων μεταφορών. Αυτή είναι μια τροπολογία της Ινές ε, ε, Γιάλα Σέντερ. Στην παράγραφο 9 θα θέλαμε να διατηρηθούν οι αναφορές που γίνονται στις νομικές πράξεις που έχουν υιοθετηθεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολλές ε, καλές προτάσεις όταν αφορά, όσον αφορά την ασφάλεια την οδική και σχετικές υποδομές για τους ευάλωτους χρήστες. Και πιστεύω πως όταν συντάσσουμε συμβιβαστικά κείμενα που καλύπτουν ε, τη 276, τη 272 και διάφορες ακόμα τροπολογίες θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την οδική ασφάλεια που είναι πολύ σημαντικό θέμα και επαναλαμβάνεται και στην Λευκή Βίβλο. Συναντηθήκαμε με τον εισηγητή, συζητήσαμε αυτά τα θέματα, του τα θίξαμε και νομίζω πως μαζί θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα με αποτέλεσμα μια πολύ καλή έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κοσμα Αλλά θα ήθελα πρώτα να καλωσορίσω ένα νέο μέλος της Επιτροπής μας που δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Είναι το μωρό της Ντανιέλα Αγιούτο. Ε, καλώς όρισε στην Επιτροπή μας. Ε, η Γιάννα πήγε καλά. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Οι πολλές τροπολογίες που υποβλήθηκαν αποτελούν όχι μόνο μια τεράστια πρόκληση για τον εισηγητή μας δείχνουν ε, ότι η Λευκή Βίβλος έχει μεγάλη σημασία παρότι δεν είναι νομοθετική πράξη. Και βέβαια δεν είναι πολύ εύκολο να συμφωνήσουμε με όλες τις τροπολογίες. Υπάρχουν όμως κάποιες που αξίζουν την υποστήριξή μας. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τι διαφορές που υπάρχουν στις υποδομές στα διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μυστικό το ότι υπάρχουν ε, πολλά μέρη της Ευρώπης που πρέπει να καλύψουν τη διαφορά. Ε, ο κομμουνισμός δεν προώθησε πολύ την ανάπτυξη σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και Ελπίζω αυτό να ληφθεί υπόψη σε κάποιες από τις τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνοχή στην Ευρώπη και η διάκριση ανάμεσα σε, παλές σε παλαιά και νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν βοηθάει. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές τροπολογίες που αναφέρονται στις ε, ίσες συνθήκες ανταγωνισμού είναι ένα θέμα που σχετίζεται με την οικονομική ανάπτυξη και τις ε, νέες θέσεις απασχόλησης στις μεταφορές. Ε, είναι κατά του προτεξιονισμού στα κράτη-μέλη που αναφέρεται ως ε, προστασία των εργαζομένων. Βλέπουμε τέτοια φαινόμενα και στον τομέα των αερομεταφορών. Στις τροπολογίες έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και θα μπορέσουμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμα Juncker. είναι υπερβολικά αισιόδοξη η Λευκή δίπλωση όσον αφορά την εκμετάλλευση των παραδοσιακών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Πάνω από το 90% του τομέα μεταφορών εξαρτάται από τα παραδοσιακά καύσιμα, κάτι που μπορεί να έχει μόνο αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Ε, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η πολιτική μιας οικονομίας απαλλαγμένης από εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα είχε αρνητικές ε, συνέπειες ε, αναφέρεται εδώ το σχιστολιθικό αέριο και θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Παύλ Τελίτσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να απολογηθώ εκ μέρους ε, της ε, συναδέλφου που δεν μπόρεσε να είναι παρούσα και μου ζήτησε να πω λίγα λόγια σχετικά με τις εξελίξεις ε, πάνω στο θέμα αυτό μέχρι τώρα. Όσον αφορά το πρώτο μέρος των συμβιβαστικών τροπολογιών, πιστεύουμε ότι είναι ισορροπημένες και ότι αντικατοπτρίζουν τον μεγάλο αριθμό των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. και προσλέπουμε στη επόμενη σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πολυτροπικότητα και η αλλαγή τρόπων μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα γίνει πιο αναλυτική συζήτηση όταν λάβουμε τη δεύτερη σειρά συμβαστικών τροπολογιών. Επιτρέψτε μου να επισημάνω κάποια σημεία στα οποία νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. Πρώτον, ε, βλέπω έλλειψη συνέπειας ε, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στα διάφορα μέσα μεταφορών. Δεύτερον, όσον αφορά την πολυτροπικότητα, θα πρέπει να μπορέσουμε να συνδυάσουμε δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους ε, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Θα πρέπει να έχουμε ιεράρχηση των προγραμμάτων που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν είμαστε πάντα συνεπείς στο θέμα, στο θέμα αυτό. Η πρώτη τελευταία παρατήρησή μου αφορά το πακέτο αερομεταφορών στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε νωρίτερα. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι μέχρι τώρα και να εξαλείψουμε τα σημεία συμφόρησης. Και τέλος, ε, έχουμε το θέμα της διαλειτουργικότητας των εθνικών ε, συστημάτων αερομεταφορών. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή. Ο εισηγητή νομίζω κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα περιμένουμε την επόμενη φάση να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Κίλεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Φαντεκάμπ για την επικοδημητική συνεργασία. Εξετάζοντας αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες, βλέπει κανείς την προσπάθεια που έχει γίνει να συνδυαστούν μεταξύ τους διάφορες τροπολογίες. Μεγάλο ερώτημα παραμένει όμως όσον αφορά τη στάση του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις COP21. Εμείς δηλαδή πώς βλέπουμε το θέμα των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών. Επίσης έχουμε το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των ορυκτών καυσίμων. Θα πρέπει να έχουμε την τόλμη να πάρουμε θέση όσον αφορά το θέμα των καυσίμων στον τομέα των μεταφορών στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε θέση. Κατά τα άλλα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Κάθε επιτυχία εύχομαι στον εισηγητή. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να καταλήξει σε καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να Ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος ε, του συναδέλφου ε, Μπασεκούτη γιατί ξέρετε όλοι κοιμήθηκε πολύ αργά και δεν μπόρεσε να έρθει. Ε, αλλά ήταν για καλό σκοπό. Σας ευχαριστώ τι, λοιπόν καταρχήν για τη συνεργασία σας κύριε Σιγητά, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη λευκή βίβλο να τοποθετηθούν οι μεταφορές μέσα σε μια οπτική βιώσιμη ε, με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, κυρίως τις ε, κλιματικές αλλαγές. Ε, οι μεταφορές δεν θα πρέπει να είναι ο πέμπτος τροχός της αμάξης και όταν μιλάμε για πρόοδο θα πρέπει να δούμε έναν οδικό χάρτη γιατί έχουμε δεσμεύσεις. Πρέπει να μειώσουμε τα αέρια του ε, θερμοκηπίου 20% ε, μέχρι το 30% και μέχρι και 60% το 2050 γιατί είμαστε μέσα σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα πλαίσιο για να μην ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς. Επίσης χρειάζεται να δείξουμε ότι οι αυριανές μεταφορές δεν θα εξαρτώνται πλέον από στερεά καύσιμα, από ορυκτά καύσιμα είναι σημαντικό λοιπόν να ε, τοποθετηθούν στους πόρους για τις ευρυνές μεταφορές αυτές οι προκλήσεις της διάρκειας, της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας. Και όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα, αυτό μας κάνει βεβαίως να μιλάμε και για την τιμή. Ε, και η τιμή εμέσως θέτει άλλο ερώτημα, φορολόγηση ή επιδοτήσεις καθώς και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με αυτό το θέμα. δηλαδή εξωτερήκευση του κόστους όπως βρίσκουμε στο πακέτο για τις οδικές μεταφορές. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε τα όσα θα ψηφίσουμε ε, ε, για τα εφαρμοστικά ζητήματα. Δεν αρκεί να έχουμε ένα λευκό βιβλίο. Πρέπει στην πράξη να έχουμε ισχυρές δράσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή και άρα να προβλέψουμε και τις νέες προκλήσεις. Είτε πρόκειται για τα θέματα που είπαμε, της ψηφιοποίησης, τα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης, τα θέματα της αποσύνδεσης των μεταφορών ανάμεσα στον ε, όγκο και την οικονομική αξία, το θέμα της ασφάλειας, τα κοινωνικά θέματα που είναι στην ατζέντα. Ο κύριος Σεκάουτ, λοιπόν, ο συνάδελφός μου, ε, σα δίνει ραντεβού για τις 2 Ιουνίου για τη δεύτερη συνεδρίαση που αφορά τι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Ευχαριστώ πολύ Πέτερ Λόντκρεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πιο σημαντικά θέματα στη Λευκή Βίβλο, κατά τη γνώμη μου, έχουν να κάνουν με το κοινωνικό dumping και με τα κεφάλαια. Στην Σουηδία ε, έχουμε μια καταστροφική κατάσταση όσον αφορά τις ε, θέσεις εργασίας. Η ε, θέσεις που, οι ε, επιχειρήσεις που προσφέρουν καλές ε, συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους τους χάνουν στον ανταγωνισμό με ξένες εταιρείε. Αυτό ονομάζεται προτεξιονισμός. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι απόλυτη περιφρόνηση των ανθρώπων που χάνουν στην κατάσταση αυτή. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα κέρδη είναι πιο σημαντικά από τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Αυτό είναι θλιβερό. Όσον αφορά την έκθεση στο σύνολό της, εξετάζουμε τις συμβαστικέ τροπολογίες, αλλά δεν ε, συμφωνούμε με όλες. Ε, το, η κοινωνική πτυχή είναι η πιο σημαντική για μας. Έχουμε επίσης ε, και την αρχή της επικουρικότητας, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της Λευκής Βίβλου θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, ε, θα έχουμε διαπραγματεύσεις για αυτές. Επίσης, ε, βιωσιμότητα, προσβασιμότητα και ψηφιοποίηση το, της αγοράς μεταφορών. Συμφωνούμε και με τις ευφυείς μεταφορές. Όπως είπα και νωρίτερα, τα σημαντικότερα για μας είναι η ασφάλεια οδηγών και επιβατών, πληροφόρηση σεβασμός του νόμου από πλευράς των επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, κάνει κάτι στον τομέα αυτών. Ίσες συνθήκες ανταγωνισμού, προστασία των κεφαλαίων και κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Νίλσεν. Ευχαριστώ πολύ. Στα σουηδικά συνεχίζω κι εγώ. Δύο θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μας. Το πρώτο αναφέρθηκε και από άλλους βουλευτές. θέματα ισότητας στον τομέα των μεταφορών. Ως δήμαρχος πριν 20 χρόνια αρχίσαμε να εξετάζουμε την ισότητα των δύο φύλων στις μεταφορές. Και βλέπω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Καλύτερες συλλογικές μεταφορές που καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. Το άλλο θέμα είναι η κοινωνική διάσταση. Πολλές τροπολογίες δικές μου και άλλων τονίζουν την, τον δίκαιο ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται εντός μιας αγοράς δεν επιτρέπεται να ε, περιφρονούν κανόνες για την ασφάλεια, για τις κοινωνικές συνθήκες, για τις συνθήκες εργασίας. Και να κερδίζουν ε, δηλαδή ε, παραβιάζοντας τον νόμο. Δίκαιες συνθήκες εργασίες και σωστές συνθήκες εργασίες είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε. Βλέπω ότι και ο Επίτροπος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Όσοι θέλουν περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς αυτής ε, μπορούν να το ξεχάσουν ε, ε, αν δεν καλύψουμε πρώτα τα κοινωνικά θέματα. Κατόπιν έχουμε το θέμα των αερομεταφορών. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις κοινωνικές πτυχές στον τομέα των αερομεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής Βάντεν Κάμπ, λευκή βίβλος δεν είναι οδηγία, δεν είναι κανονισμός. Θα θυμάστε ότι η λευκή βίβλος πριν από 11 χρόνια ήταν ένα στιγμιότυπο εκείνης της εποχής. Και από τότε κάποια όνειρα εκπληρώθηκαν κάποια άλλα που δεν εκπληρώθηκαν. Είναι μια συγκέντρωση ιδεών αυτό, μια συλλογή ιδεών. Και ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές θα συμβάλλουν στο να κάνουμε την απεικόνηση της στιγμής, να διαγνώσκουμε, να διαγνώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για τις τροπολογίες. Δεν θα επεκταθώ γιατί δεν θα με αφήσει ο Πρόεδρος να σας πω ότι δεν είμαι δογματικός ε, ως προς τις τροπολογίες. Θέλω να είναι συμβατές με τη γενικότερη μας πρόθεση. Ε, βέβαια, εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες που τις θεωρώ τις πιο κατάλληλες και σκόπιμες. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο δεν είναι ρεαλιστική να ως ε, Εννοώ δηλαδή ότι η πλήρης ανεξαρτησία δεν είναι κάτι το ρεαλιστικό. Μπορεί να μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο, αλλά όχι να ε, εξουδετερωθεί πλήρω να μειωθεί στο μηδέν. Και πρέπει να τονίσουμε την συμπλήρωση των διασυνοριακών υποδομών. Η ακόμα μεγαλύτερη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Και είναι απαραίτητο να αναφέρουμε την εδαφική συνοχή πάντοτε κάθε πολιτική πρέπει να τη λαμβάνει υπόψη της στην εδαφική συνοχή ε, βάσει της συνθήκης. Ισορροπία των τρόπων μεταφορών, πολυτροπικότητα. Είναι πολύ σωστό. Ωστόσο οι μεταφορές από τον αυτοκινητόδρομο είναι προϊόν βολονταρισμού. Δηλαδή, μπορεί να θέλουμε να προωθήσουμε και άλλου τρόπου, αλλά εν πάση περιπτώσει οι μεταφορέ μέσω αυτοκινητόδρομων με φορτηγά υπάρχουν σήμερα, δεν μπορούμε να τι παραμερίσουμε. Πρέπει να δούμε και το θέμα των λιμένων. Και πρέπει να δούμε πώς ελήφθησαν αποφάσεις που θεωρούνται σωστές στην εποχή και σήμερα πλέον θεωρούνται ανεδαφικές ή εξωφρενικές, ειδικά σε σχέση με την περιοχή των Άλπαιων. Και πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ε, ε, το, την σύγχρονη σκέψη και την αποτελεσματικότητα. Αυτές είναι οι προσταγές μας. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθεια που κατέβαλε. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες όλων των τροπολογιών που έχουμε υποβάλει, 37 το σύνολο. Θέλω όμως να πω ότι ως προς αυτή τη λευκή βίβλο συμφωνούμε ότι περιλαμβάνει ή δεν περιλαμβάνει κάποιες λεπτομέρειε καλός ή κακός, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίζει. Πρώτον, να κάνει διάγνωση για τα προβλήματα. Ποια απεικόνηση των προβλημάτων, ποια προβλήματα υπάρχουν, ποια προβλήματα είχαμε ω κοινοβούλιο με την προηγούμενη λευκή βίβλο. Ο κορεσμός στην Ευρώπη μα στοιχίζει μία ποσοστιαία μονάδα του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ένα μόνο νούμερο σας δίνω και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Ο κορεσμός με την έννοια ότι έχουν εξαντληθεί τα μέσα μεταφορών. Δεύτερον, συνοχή να απαιτήσουμε όλα να συνάδουν με τις οδηγίες και τους κανονισμούς που συμπληρώνονται και εγκρίνονται με συστηματικό τρόπο. Επομένως, σε όλα τα θέματα που συζητούνται, σε όλες τις επιτροπές, σε όλες τις συνεδριάσεις, για όλες τις εκθέσεις, πρέπει να υπάρχει συνοχή με αυτό που προβλέπεται στις οδηγίες, με, αυτό που προβλέπονται που προβλέπεται στα έργα για τα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα και πρέπει με αποφασιστικό τρόπο επιτέλους να προσεγγίσουμε το θέμα του ενιαίου ουρανού, Single Sky. Πρέπει να δούμε το δίκτυο του Γαλιλαίου, να οριστικοποιηθεί αυτό το έργο, να τελειώσει πια. Η Επίτροπος πριν από δύο εβδομάδες πριν από δύο εβδομάδες παρουσίασε 16 πρωτοβουλίες για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεκίσουμε επιτέλους την ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά. Επομένως οι εκθέσεις και τα project, τα διάφορα έργα δεν είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Να υπάρχει συνοχή, συνεκτικότητα και με το τέταρτο, ε, την τέταρτη δέσμη μέτρων για τα σιδηροδρομικά. Το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο που ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε τους επόμενους μήνες μεταξύ άλλων. Είπατε ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ε, πολλοί περιορίζονται μόνο να σχολιάσουν τις δαπάνες και όχι τα έσοδα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν έσοδα για να εκτελέσει κανείς ένα έργο. Πρέπει να αξιοποιήσει σωστά και καλά τους πόρους. Και τι έχουμε δει μέχρι τώρα ότι έχει υπάρξει χρήμα που έχει κινηθεί στα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη το χρησιμοποίησαν με τραγικό τρόπο, γιατί δεν έδωσαν προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά έργα. Άρα περισσότερη συνοχή στις απαιτήσει ως προς τα έξοδα και τις δαπάνες. Και για λόγους συνοχής, και συνεκτικότητες πρέπει να τονίσουμε το στρατηγικό ρόλο της βιομηχανίας για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης επιτέλους και στη Λευκή Βίβλο να μιλήσουμε επιτέλους για την τροπικότητα ή την πολυτροπικότητα που αναφέρει ο συγητής, συμφωνούμε εδώ απολύτως. Ωστόσο, το κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής, να μιλήσουμε ξεκάθαρα για αυτούς τους κλάδους και για άλλους. Συγκεκριμένοι πόροι για καινοτομία, για έρευνα. Shift to rail. Πώς θα κάνουμε αυτό το δικό μας κοινό εγχείρημα του να μεταστραφούμε και να ε, προσχωρήσουμε και να προσεγγίσουμε περισσότερο το σιδηρόδρομο. Ο εισηγητής δεν αναφέρθηκε στην ανάγκη σε όλη αυτή τη βίβλο ε, τη Λευκή Βίβλο να ξεκαθαρίζουμε το ότι η πολυτροπικότητα, η έρευνα, η καινοτομία πρέπει να είναι πράγματα καλά προσαρμοσμένα και προσβάσιμα για όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες και για όλους τους ανθρώπους που ε, παρουσιάζουν μειωμένη κινητικότητα. Άρα πληροφόρηση, ενημέρωση, επόμενο κεφάλαιο. Αν κάνουμε τα, πράγματα σωστά, οι νέε θέσει απασχόληση που θα δημιουργηθούν χρειάζονται να έχουν ενημερωθεί άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο. Να έχουν ενημερωθεί για τον έξυπνο τρόπο μεταφορά, για τι έξυπνε μεταφορέ. Ένα κεφάλαιο στη βίβλο πρέπει να το αφιερώσουμε εκεί, στι αναδιαρθρώσει που πρέπει να γίνουν εάν τελικά εκτελέσουμε και εφαρμόσουμε αυτό το έργο με συνοχή και να ενημερώσουμε τους ανθρώπους και να τους καταρτήσουμε στην Ευρώπη με εναρμονισμένο τρόπο, με συγκεκριμένα κριτήρια, γιατί αυτό θα διευκολύνει την κοινωτικότητα των Ευρωπαίων. Και τέλος, διαφάνεια. Πρέπει να απαιτήσουμε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφάνεια τρεις φορές στη χρηματοδότηση των έργων και στις διαδικασίες απλούστευσης. Και τελικά να σας πω και το εξή. Έχουν σημασία οι λεπτομέρειες και θα σας πω για μία και μόνη τροπή τροπολογία, την 249. Η πρόταση της Κομισιόν υπογραμμίζει ότι οι κινητήρες των οχημάτων των δίτροχων και εγώ υπέβαλα τροπολογία αυτό να αλλάξει και να γίνει τρίτροχων. Γιατί, γιατί στην προηγούμενη θητεία είχαμε μια καινοτόμα επιχείρηση νέων ανθρώπων που έφτιαξαν ένα συνεταιρισμό και είχαν ένα project, ένα έργο τρίτροχου τρίτροχου οχήματος για να διευκολύνουν ακριβώς αυτούς τους πολίτες που δεν μπορούσαν να υπεύσουν δίτροχο όχημα. Και γιατί δεν μπορούσαν, γιατί δεν τους επέτρεπε ο κανονισμός να βγάλουν δίπλωμα για μηχανή ε, δίτροχη. Και επομένως η εταιρεία αυτή έφτιαξε τρίτροχο για τέτοιου είδους άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Και είναι μια εξαιρετική καινοτομία αυτή, γιατί να μην μπορούν να ε, βγάλουν τέτοιο δίπλωμα. Ε, επομένως γι' αυτό έκανε αυτή την τροπολογία πάντοτε με ορίζοντα την καινοτομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κριστίνη Βουταλό. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για το σπουδαίο έργο που ξεκίνησαν και που θα χρειαστεί να συνεχίσουν να κάνουν. Κατανοώ και ότι 600 ε, και άνω τροπολογίες είναι τεράστια δουλειά για την εξέβριση συμβαστικών. Ωστόσο, ταυτόχρονα δείχνει και την ζωτικότητα και τη δυναμικότητα των Ευρωβουλευτών για να προχωρήσουμε και για να υποβάλλουμε σοβαρές προτάσεις όσον αφορά τις προπτικές της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών. Και ήθελα να επιμείνω για κάποιες από τις πολλές τροπολογίες που υποβάλαμε, συχνά ομαδικά, Ιδιαίτερα στο θέμα που αφορά την πλαισίωση, δηλαδή το να έχουμε μια πραγματικά εναρμονισμένη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαμε συζητήσει παλιότερα τα θέματα της χρηματοδότησης ε, του σχεδίου ΕΦΣΥ είναι σημαντική λοιπόν αυτή η περίπτωση και στηρίζουμε και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κοστολόγηση των ε, οδικών υποδομών. Θα πρέπει όλα αυτά λοιπόν να αναλυθούν υπόψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης έχουμε την τροπολογία όπου ζητούμε τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου ταμείου για τη χρηματοδότηση των δημοσίων μεταφορών. Καταλάβουμε πολύ καλά και η προηγούμενη αμέσως συζήτηση μας παραπέμπει σε αυτή τη διάσταση που πρέπει επίσης να έχει το, τη θέση της στην ανθεώρηση του Λευκού Βιβλίου για τις μεταφορές. Να τονίσω επίσης τις τροπολογίες που θα νομίζω θα περιλαμβάνονται μόνο στι συμβιβαστικέ όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα για τα ελαφριά και για τα βαριά οχήματα μετά το 2020 και να θυμίσω επίσης ε, το στόχο μείωση 30% του διεξιδίου του άνθρακα για τι συνδυασμένε μεταφορέ μέχρι το 2030 στην πρόταση του Λευκού Βιβλίου. Οι νομοθετικέ προτάσει που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ε, μέσα στο, για την εφαρμογή του πακέτου κλίμα και ενέργεια θα πρέπει να τηρούν αυτέ τι προδιαγραφέ. Επίση, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη τι προτάσει κλειδιά, όπω η διπλασιασμό τη ε, ε, χρήσης των δημοσίων μεταφορών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, αναφέρθηκε στην ε, πεζή κυκλοφορία. Θα ήθελα όμως να πω γιατί είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχουν ε, οι δρόμοι Eurovelo και δεν γνωρίζω ούτε μία που να περνάει από τους δρόμους ε, για να λειτουργήσουν καλά θα πρέπει να περνάνε μέσα από τις πόλεις. Έχουμε για παράδειγμα ποδηλατόδρομο στο Βερολίνο που επιδοτείται από την Ευρώπη και από την ε, Γερμανία. Ε, και όσον αφορά την πεζή κυκλοφορία δεν γνωρίζω κανένα μέσο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να περπατήσει κανείς. Θα πρέπει να περπατήσει κανείς μέχρι το αυτοκίνητό του για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών και στις πόλεις και δεν μπορούμε να το παραμελήσουμε. Και ευχαρίστω σας αναφέρω το παράδειγμα της Κοπεχάγης. Εάν κάποιος έλεγε πριν 20 χρόνια ότι πάνω από το μισό των ανθρώπων στην Κοπεχάγη θα πηγαίνανε στη δουλειά με ε, το ποδήλατο ή με τα πόδια, θα λέγανε μα ονειρεύεσαι. Και όμως ε, σήμερα το 53% των ανθρώπων έτσι πηγαίνει στη δουλειά του ή στο σχολείο. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως. Ε, στη, στο Βερολίνο έχουμε χτίσει αυτοκινητόδρομο που θεωρείται αυτοκινητόδρομος και τώρα μόλις ακούω ότι το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ε, θα χρηματοδοτηθεί ε, περιφερειακός αυτοκινητόδρομος ε, των Βρυξελών. Αυτό αφορά αποκλειστικά την πόλη, δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Όταν όμως μιλάμε για το ποδήλατο λέμε «Α, όχι, απεικουρικότητα» κλπ. Να σας αναφέρω άλλο ένα στοιχείο. Ο τουρισμός με ποδήλατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 44 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Το ίδιο με τα κρουαζιερόπλια. Εάν μια πόλη πει ότι α, πρέπει να φροντίσουμε το λιμάνι μας, ε, χρειάζομαι 2 δισεκατομμύρια για τα κρουαζιερόπλια, δεν ε, υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως κάποιος ζητήσει 2 δισεκατομμύρια για ε, τους ποδηλάτες, θα θεωρηθεί αυτό υπερβολικό. Παρακαλώ λοιπόν να ε, σκεφτεί Βήμ να το συμπεριλάβεις αυτό στην ε, έκθεσή σου, διότι δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν. Ξέρω ότι τα αυτοκίνητα θα είναι απαραίτητα και στο μέλλον, αλλά και τα άλλα στοιχεία θα είναι απαραίτητα και γι' αυτό δεν πρέπει να αποκλείσουμε κανέναν τρόπο μεταφοράς. Παρακαλώ να ακολουθήσεις αυτή μου την παρατήρηση. Ε, η Κομισιόν τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν ε, θα αναφερθώ στην ποδηλασία, θα το εξετάσει αυτό ε, η συναδελφός μου όσον αφορά το περιβάλλον. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι για την έκθεση αυτή. Είναι πολύ καλή η δουλειά που έχει γίνει. Και το χρονοδιάγραμμα είναι ιδανικό. Παρακαλώ λοιπόν να το τηρήσετε. Οι τροπολογίες όπως τόνισαν αρκετοί από εσά ε, δείχνουν όχι μόνο την δημιουργικότητα της Επιτροπής σας αλλά και την αφοσίωσή σας ε, στην βιωσιμότητα στις μεταφορές και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για την εκπόνηση συμβαστικών τροπολογιών. Ε, πάντως παίρνουμε πολύ στα σοβαρά όλο το υλικό αυτό κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, εν ώψη της επόμενης συνεδρίασής σας στις 2 Ιουνίου όπου θα εξετάσετε τη δεύτερη σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να στείλετε σαφές μήνυμα όσον αφορά την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Αυτό το έχω πει επανειλημμένα, είναι ευαίσθητο και πολύ σημαντικό θέμα. Χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική υποστήριξη όσον αφορά τις οδικές μεταφορές. Παρακαλώ μην θεωρήσετε ότι οι οδικές μεταφορές αντίκυνται, ε, είναι κάτι αντίθετο, διαφορετικό από τα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ότι αποτελούν πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε όλοι ότι η αγορά μπορεί να συνδυάζεται με κοινωνικές ρυθμίσεις και μπορούμε έτσι να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε την ποιότητα των συνθήκων εργασίας στον σημαντικό αυτόν τομέα. Επίσης έχουμε το θέμα του οργανισμού. Το θέμα μας ε, δεν είναι ε, απαραίτητα ένας νέος οργανισμός, ούτε θέλουμε να αποκτήσουμε νέες ε, εξουσίες, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν καλύτερη δουλειά όσον αφορά την εφαρμογή, τον προγραμματισμό για να οργανώσουν ε, έναν καλό και αποτελεσματικό τομέα οδικών μεταφορών. Τρίτον, λιμάνια. Το θέμα των ε, λιμανιών δεν είναι μόνο θέμα ρύθμισης. Ξέρω ότι δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός όσον αφορά ε, την σχετική οδηγία, αλλά υπάρχουν πολλές σημαντικές στοιχές που συνδέονται με τους λιμένες. Ακούσαμε κάποιες πρωτότυπες ιδέες. Έχετε καταφέρει να βάλετε τα λιμάνια στο κέντρο των διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, θα πρέπει να το σκεφτείτε όμως και εδώ πέρα. Και όσον αφορά τις αστικές μεταφορές, είναι πολύ σημαντικές και είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε όλοι αυτόν τον ε, σκόπελο της επικουρικότητας. Το θέμα δεν είναι αν παραβιάζεται η επικουρικότητα, το θέμα είναι να διασφαλίσουμε σε όλες μας τις εργασίες να λαμβάνουμε υπόψη τις συνέπειες και να εξετάζουμε τι θα είναι χρήσιμο για τις πόλεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να απλοποιήσουμε και να συνδυάσουμε τις πολιτικές μας και για το αστικό περιβάλλον. Και εδώ είστε πρωτοπόροι όσον αφορά την ένταξη της αστικής διάστασης στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτές αυτή την προσέγγιση. Τέλος, όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Αρκετοί από εσά αναφέρθηκαν στο ψηφιακό θεματολόγιο. Και εδώ χρειάζομαστε τη βοήθειά σας. Θα πρέπει να καθορίσετε σημαντικές προτεραιότητες όσον αφορά αυτά που απομένουν να γίνουν. Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της διαλειτουργικότητας, κάτι που πολύ σοφά ανέφεραν κάποιοι από εσά και θα πρέπει να μάθουμε πώς να ανταποκρινόμαστε σε νέες προκλήσεις όπως είναι η μοιρασμένη οικονομία και οι συλλογικές μεταφορές. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό υπό το φως της χρήσης της νέας τεχνολογίας και όχι άλλες στοιχείες. Και τέλος, το θέμα της ψηφιοποίησης έχει να κάνει και με την πρόσβαση σε δεδομένα. Χρειαζόμαστε πολύ υποστήριξη από σας στο θέμα αυτό, διότι υπάρχει σημαντική αντίθεση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς του τομέα μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Βιμ Φαντεκάμπ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για αυτές τις πολύτιμες ε, παρεμβάσεις. Θα πρέπει να σας πω πως ε, γίνονται ε, παρατηρήσεις ε, για τις συμβαστικές τροπολογίες που δεν μπορείτε να έχετε δει ακόμα γιατί τις συζητήσαμε μόλις χθες το απόγευμα. Αλλά φαίνεται να γνωρίζουν ήδη τι θα υπάρχει μέσα σε αυτές τις ε, συμβαστικές. Δεν έχουμε όμως ολοκληρώσει τη συζήτηση, γι' αυτό αυτό έχει ελκύσει την προσοχή μου. Αυτό σημαίνει πως έχουμε Καλέ επαφέ όσον αφορά το ποδήλατο και το περπάτημα. Συμφωνώ πως είναι ένα θέμα αρχής και αν ήταν μια παρατήρηση η επίκριση είναι θετική επίκριση. Εγώ όταν δεν χρειάζεται να πάρω το αυτοκίνητό μου περπατώ. Αλλά είναι η Ευρώπη που πρέπει να μου πει πότε και πού θα πρέπει να περπατήσω. Είναι ένα θέμα αυτό. Και επίσης, η κυκλοφορία στις Βρυξέλλες. Δεν θα πρέπει να είναι το σημείο κίνησης, γιατί είναι πολύ λυπηρή η κατάσταση. Οι αυτοκινητόδρομοι φτάνουν μέχρι το παλάτι σχεδόν. Είναι μια τρέλα. Αλλά όταν μιλάμε για διπλασιασμό της προσφοράς ε, των δημοσίων μεταφορών εντός των πόλεων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αν πρέπει όμως να δούμε το περπάτημα και το ποδήλατο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Σε τουριστικό επίπεδο είναι πολύ όμορφο, εντάξει, αλλά Καλύτερα είναι να συγκεντρώσουμε τροπο, τρο, συμβιβαστικές τροπολογίες ε, ε, και χάρη ε, και μάλλον θα σας ενημερώσουμε ανάλογα με τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές και να ευχηθώ κάθε επιτυχία. περνάμε τώρα το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Η συγγήτρια είναι η Καρή Μαντελή, της δίνω το λόγο. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν γίνεται λόγος για κινητικότητα πρέπει να υποθεί ότι η κινητικότητα δεν είναι αυτός σκοπός λογικά και φυσιολογικά η κινητικότητα θα πρέπει να είναι δικαίωμα για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Το 85% των Ευρωπαίων πολιτών θα ζουν σε πόλεις, λίγαν συντόμως. Και άρα η κινητική η κινητικότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε πόλεις όλων, ε, ακόμα και για τα άτομα μειωμένη κινητικότητα. Ενθάρρυνση της πρόσβαση στο σχολείο, στον πολιτισμό, στου χώρου ψυχαγωγία στους χώρους εργασίας. Ωστόσο, σήμερα η αστική κινητικότητα είναι περιοριστική. Η εξάρτηση από τα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα η κυκλοφοριακή συμφόρηση κάνουν τους πολίτες ε, ε, ε, να είναι εγκλωβισμένοι όχι στην κινητικότητα που επιλέγουν, αλλά στην κινητικότητα που υφίστανται. Και φτάνουμε στα όρια του παραλόγου, στο βαθμό που το 50% της μετακίνησης μέσα στο αστί δεν ξεπερνά την απόσταση των 5 χιλιόμετρων. Επομένως, φιλοδοξία της έκθεσης είναι να επαναπροσανατολίσει την αστική κινητικότητα προς τρόπους μεταφοράς βιώσιμους με σκοπό να ανταπεξέλθει στις διάφορες προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας τον 21ο αιώνα. Πρώτον, την κλιματική αλλαγή. Η γεωργία και η βιομηχανία έχουν μειώσει τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως οι μεταφορές το έχουν αυξήσει κατά 30%. Ε, η κυκλοφορία η είναι αυτή που εφείλεται για το 1 τέταρτο της, α, των, της αύξησης των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και έχουμε το στόχο ε, μείωσης κατά 30% με ορίζοντα το 2030. Δεύτερη μεγάλη πρόκληση, η υγειονομική. Οι μεγάλες πόλεις ζουν με ρήπους που εκτοξεύονται. Κάθε χρόνο 400.000 πρόοροι θάνατοι οφείλονται στα πολύ λεπτά ε, σωματίδια που εκπέμπονται από τις εξατμίσεις των κινητήρων diesel. Θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η ρήπανση από, το, από τα αυτοκίνητα θα είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας παντού στον κόσμο, βάσει της μελέτης του ΟΗΕ. Θα πρέπει να προλάβουμε και να προβλέψουμε. Τρίτη μεγάλη πρόκληση, το επίγον. Ο επίγον χαρακτήρας ως προς τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου. Οι χρήστες των αυτοκινητόδρομων ε, βρίσκονται σε κίνδυνο. Το 38% των θανάτων οφείλεται ε, σε το ε, θανάτων που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα είναι ατυχήματα που έχουν σημειωθεί μέσα στις πόλεις. Πάρα πολλοί πολίτες αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους και των εισοδημάτων τους στις μεταφορές και ορισμένοι δεν έχουν πρόσβαση κιόλα στις μεταφορές. Ένα παράδειγμα, στη δική μου χώρα, στη Γαλλία. 8 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην βιώσιμη κινητικότητα, ούτε καν στην αστική κινητικότητα. 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Άρα δημιουργούμε ένα νέο φαινόμενο. Είχαμε ενεργειακή αβεβαιότητα με τις πηγές ενέργειας και τώρα θα έχουμε ε, αβεβαιότητα ως προς την κινητικότητα. Και πρέπει αυτά να τα προλάβουμε και να τα προβλέψουμε. Υπάρχει άλλη κινητικότητα και είναι αυτή απαραίτητη. Όλοι οι τρόποι μεταφορέας να εξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη την αηφόρο, τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να ερευνάτε συνεχώς το σημείο ισορροπίας μεταξύ του αντικτύπου των μεταφορών στο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, ούτω καθεξής. Πρέπει να βρίσκεται το σημείο ε, ε, ισορροπίας μεταξύ των αναγκών των σημερινών ανθρώπων και της επόμενης ε, γενεάς. Στον 21ο αιώνα μπορούμε να κάνουμε προοπτικές επιτέλους μελέτες και όχι να λειτουργούμε πυροσβεστικά, όχι να λειτουργούμε κοντόφθαλμα με ορίζοντα 5-10 ετών, αλλά αντίθετα σε βάθος χρόνου, με οραματική θεώρηση, σε βάθος 20-30 και πλέον χρόνων. Τις παραμονές της Συνόδου Κορυφής για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η ενεργειακή ασφάλεια να, και αποδοτικότητα να είναι στο επίπεδο επίκεντρο της αστικής κινητικότητας είναι κάτι που το θέλει και η τοπική αυτοδιοίκηση και γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν τη συγγραφή ενός νομοθετικού πακέτου με τίτλο «Κλίμα και μεταφορές» για να προσδιορίσει συγκεκριμένους στόχους ε, δεσμευτικούς για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τα μέσα μεταφοράς. Θα μπορούσε η Κομισιόν να ε, ε, εξαλείψει το ντίζελ από τα αστικά κέντρα μέχρι το 2020 και τελικά να εξαλειφθούν πλήρως μέχρι το 2050. Αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πρημοδοτήσουν ε, καύσιμα μη ορυκτά μορφές ενέργειας που δεν θα είναι ορυκτά καύσιμα όσο το περισσότερο για να ε, τροφοδοτήσουν και να θέσουν σε κίνηση τα συστήματα μεταφορών. Ερχόμαστε τώρα στους ίδιους τρόπους μεταφοράς. Ε, το τελεφερίκ, το τραμ, ε, το, το μοίρασμα του αυτοκινήτου κατά το οποίο ένας εργαζόμενος με αυτοκίνητο παίρνει και άλλους εργαζόμενους μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο για να μεταβεί στο χώρο εργασίας τότε Ελευθερίκ μεταξύ άλλων, όλα αυτά είναι μέσα που θα πρέπει να ε, καταγραφούν και να ενθαρρυνθούν. Δεν έχουν όλα τα κρατη ούτε όλες οι τοπικές και περιφερειακές αρχές σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκαταστήσει αυτό το κενό, ε, επιβάλλοντας ε, τα η χρηματοδότηση για την αστική κινητικότητα να εξαρτάται από το κατά πόσο οι τοπικές αρχές ή το εθνικό κράτος έχει εσωτερνιστεί και έχει συντάξει σχέδιο βιώσιμη κινητικότητα. Τα σχέδια αυτά είναι μοχλή δράσης για να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωση για τη μείωση των εκπομπών αερίων ε, φαινομένου θερμοκηπίου αλλά και για τη μείωση των ατυχημάτων. Ένα προβληματισμό σε περισσότερο βάθο θα αναδειχθεί στην έκθεση αυτή. Γίνεται λόγος για τη ταχύτητα και για τις υπερβάσεις. Καλό τα κράτη-μέλη και τις τοπικές αρχές να επιβάλλουν όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην πόλη έτσι ώστε να ε, με ορίζοντα το 2020 το 2013 για να ε, συνάδουν τα οχήματα με τους άλλους τους πιο ήπιους τρόπους μεταφοράς. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι το τελευταίο χιλιόμετρο παράδοσης είναι πολύ σημαντικό. Ε, εκεί είναι που δημιουργείται περισσότερη ρύθμιση, ε, ε, ρήπανση, με συγχωρείτε. Επομένως, όταν τα logistics, η επιμελητή, ο εφοδιασμός γίνεται με, έναν οικολογικό τρόπο για το τελευταίο χιλιόμετρο της παράδοσης των αγαθών, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και... Για να υλοποιήσουμε την ε, βιώσιμη αστική κινητικότητα πρέπει να κάνουμε επενδύσεις το όνομα των επενδύσεων θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Η κινητικότητα έχει ανάγκη, χρειάζεται ποιοτικέ επενδύσεις γιατί είναι υπηρεσία κοινή ωφελία, δημοσίου συμφέροντος. Έχουμε πάρα πολλές υποδομές απαξιωμένες και δαπανηρές προτείνω 50% των εσόδων από την Ευρωβινιέτα να δοθούν σε project βελτίωσης της αστικής κινητικότητας. Το 75% των διοδίων για το κλινόν άστη να δοθούν σε βελτίωση της κινητικότητας ε, στις πόλεις και αυτό θα πρέπει να το υπερασπιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω του ΦΕΝΤΕΡ μαζί με το Ταμείο Συνοχής όπου υπάρχουν προγράμματα για την βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις στρατηγικές επενδύσεις σε σχέδια έρευνας και καινοτομίας που έχουν σχέση με τις αστικές μεταφορές και είμαι ευτυχής που σήμερα το πρωί άκουσα ότι στο πλάνο Juncker, σχέδιο Juncker υπάρχει αυτό το στοιχείο και ευχαριστώ τους εισηγητές που αγωνίστηκαν για την ανάπτυξη της ε, ε, πολιτικής για τις πόλεις. Είναι μια έκθεση που ε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό θέμα για αυτή τη θητεία ε, θα μας επιτρέψει να συμφιλειωθούμε με τους ε, ε, συμπολίτες μας. Είναι θέματα πολύ συγκεκριμένα, πολύ απτό και με τους συνσηγητές της Σκιώδης θέλω να τους ευχαριστήσω για την συνεργασία τους σε αυτά τα σημεία έχουμε καταλήξει. Βεβαίω η συνεργασία μας θα συνεχιστεί στις επόμενε εβδομάδε, γιατί το μήνυμα είναι να δώσουμε μια έκθεση η οποία δεν θα είναι μόνο στο ύψος των προσδοκιών και των αναγκών των που έχουν εκφράσει οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Εγώ θέλω να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και των πολιτών. Σα ευχαριστώ λοιπόν ε, από τον Πορτέρα για τα σχόλιά σα και για τι προτάσει σα. Ευχαριστώ πολύ. Κλάουδια Σμίτ, Ιζαμπέλα Τεμόντε, Λουκασέφσκα, Τίτερ Κόχ. Ωραία. Ωραία, κλείνουμε το κατάλογο των ομιλητών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ανέφερε και η εισηγήτρια, η αστικοποίηση αποτελεί παγκόσμια τάση που κάνει την ε, κινητικότητα όλο και πιο σημαντικό θέμα. Ήδη έχουμε συνεργαστεί με την εισηγήτρια ε, και πριν αυτό το σχέδιο έκθεσης αλλά πρέπει να πω ότι δεν βλέπω τη συνεισφορά της δικής μου πολιτικής ομάδας στο σχέδιο έκθεσης και υπάρχουν κάποια θέματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω, όπως είναι η δυνατότητα παροχής ε, δωρεάν συλλογικών μεταφορών ή η απαγόρευση των αυτοκινήτων στις πόλεις. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά όλοι να συμφωνήσουμε ε, με το τελικό σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα να θίξω τρία θέματα που θα ήθελα να δω στην τελική έκθεση. Καταρχάς τον ρόλο της, του αστικού σχεδιασμού. Ελπίζαμε ότι τα χωροταξικά θέματα θα τονίζονταν περισσότερα στην έκθεση αυτή. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η πιο σημαντική φράση για να δημιουργήσουμε ε, δίκτυα ομαλών και αποτελεσματικών υπηρεσιών. Ξέρουμε ότι οι σχετικές αποφάσεις ε, έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες ε, όσον αφορά την κυκλοφορία, την ασφάλεια και τους διάφορους τρόπους μεταφορά. Η συγγήτρια τονίζει το ρόλο της πεζοπορίας και της ποτηλασίας. Ξέρουμε ότι αν αυτά ληφθούν υπόψη εγκαίρως, είναι πιο πιθανό να ε, αποτελέσουν πραγματική δυνατότητα επιλογής ε, για τους ε, χρήστες. Σημαντικό όμως είναι να μην ξεχάσουμε τα αυτοκίνητα, διότι συνεχίζουμε να χρειαζόμαστε αυτοκίνητα στις πόλεις και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι οι ευφυείς και καινοτόμες τεχνολογίες. Με καινοτόμε λύσεις, οι μεταφορές θα είναι πιο αποτελεσματικέ, ασφαλεί και πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Οι επιβάτε θα λαμβάνουν πληροφορίε σε πραγματικό χρόνο για τις ε, συνθήκες και θα χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά οι υποδομές. Τα προβλήματα κινητικότητε ε, δεν λύνονται με νέες υποδομές. Χρειαζόμαστε νέες υποδομές, είναι σημαντικό όμω επίσης να χρησιμοποιήσουμε πιο σοφά τις υπάρχουσες υποδομές. Αυτός ο στόχος θα απαιτήσει στενή συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους ε, ενδιαφερόμενους, ε, ε, τη χρήση διαφόρων λύσεων και την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών όλοι οι τρόποι μεταφορών θα πρέπει να επικεντρωθούν στην χαμηλή κατανάλωση καυσίμων. Είναι όμως σημαντικό αυτό να το προσεγγίσουμε με τρόπο ουδέτερο όσον αφορά την τεχνολογία. Δεν θα πρέπει δηλαδή να τονίσουμε κάποιες λύσεις, διότι έχουμε ήδη κάποιες δυνατότητες χρήσης ε, καυσίμων χαμηλών σε εκπομπές. Όσον αφορά τις καινοτόμες ε, λύσεις κινητικότητας και την ψηφιοποίηση, που μπορεί να δώσει πολλές νέες δυνατότητες στον τομέα των μεταφορών. Απαιτείται οι χρήστες ε, να αναλάβουν πιο προορατικό ρόλο και τίθεται και το θέμα των δεδομένων στις, μεταφορά, στις μεταφορές. Έτσι θα δημιουργηθεί η απαραίτητη πλατφόρμα για την κινητικότητα. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε τον ρόλο της ψηφιοποίησης στις μεταφορές, διότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες στον τομέα αυτών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγήτρια, ήθελα να θίξω τα θέματα αυτά αυτή τη στιγμή και θα υποβάλουμε διάφορες τροπολογίες. Ελπίζουμε μετά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια κοινή λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους ε, εργάστηκαν πάνω στην έκθεση αυτή. Ήταν εξαιρετική εμπειρία η συνεργασία με την Καρίμα Αντελή και με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές και με τους συναδέλφους μου ε, από τους σοσιαλδημοκράτες πάνω στην έκθεση αυτή. Και κατάλαβα πόσο τονίζει η Επιτροπή μας το να γίνει κάτι σοβαρό όσον αφορά την αστική κινητικότητα, διότι είναι ένα θέμα που συζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι η Καρίμα έχει απόλυτο δίκιο που τονίζει το θέμα κλειδί της επενδύσεις και το μεγάλο χάσμα επενδύσεων που υπάρχει στον τομέα αυτών. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντική πτυχή για μας. Οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ακριβώς πόσο σημαντικό είναι αυτό και όταν μιλάμε για ε, χάσμα 25 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όλη την Ευρώπη, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι και η συζήτηση που είχαμε πριν για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι πάνω από το 80% των ανθρώπων θα ζουν στο μέλλον σε πόλεις και ξέρουμε επίσης τα προβλήματα, γνωρίζουμε τα προβλήματα αλλαγής του κλίματος που τόνισε και η συγκήτρια. Αυξάνονται οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές. Προδεύουμε σε άλλους τομείς, όχι όμως εδώ. Και μεγάλο μέρος των εκπομπών προέρχεται από τις αστικές μεταφορές. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να αγνοήσουμε την κατάσταση στις πόλεις. Ε, Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αλλαγή του κλίματος και το θέμα αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων ε, και της ρήπανσης. Επίσης ε, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις πτυχές της υγείας και επικροτούμε το γεγονός ότι αναφέρονται και αυτές. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση. Έχουμε και άλλα θέματα, την ασφάλεια στους ε, δρόμους, τα δικαιώματα των πεζών, τα άτομα με αναπηρίες. Συμφωνούμε με την γενική προσέγγιση να δώσουμε προτεραιότητα στους πεζούς και στους ποδηλάτες, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την διατύπωση στην έκθεση. Και θέλουμε η έκθεση να ενισχυθεί όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Και πάλι η απόλυτη απαγόρευση μπορεί να μην αποτελεί τη λύση. Το 73% των Ευρωπαίων πολιτών λένε ότι η, ασφάλεια, η οδική ασφάλεια είναι πρόβλημα στις πόλεις. Το ότι μοιράζονται τους δρόμους μεγάλα οχήματα ή γενικά τα οχήματα με τους πεζούς και ποδηλάτες ε, καθιστά επικίνδυνους στους δρόμους. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να γνωρίσουμε στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Από πλευράς σοσιαλδημοκρατών θα υποβάλλουμε εκθέσεις για τις θέσεις απασχόλησης, ε, την ε, κοινωνική ένταξη και τον κοινωνικό διάλογο. Θα πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε τις ε, επιρροές των μεταφορών στις θέσεις απασχόλησης. 1,2 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης συνδέονται με τις αστικές δημόσιες μεταφορές ε, και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την κοινωνική διάσταση όπως ανέφερε η Κλάουδια. Συμφωνώ με το θέμα της χωροταξίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για έκθεση αστικής κινητικότητας. Συμφωνώ και με το θέμα των ευφυών τεχνολογιών, αλλά δεν θα πρέπει να γελιόμαστε. Η ευφυής τεχνολογία δεν είναι απάντηση σε όλα. Ε, χωρίς τον ε, σωστό προγραμματισμό δεν ε, θα μπορέσει να αποτελέσει την κατάλληλη λύση. Και επίσης, η Όσον αφορά την εφοδιαστική, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να είναι βιώσιμος αυτός ο τομέας. Και όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες είναι κρίσιμη σημασία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πόλεις μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Ε, στα βόρεια, τα νότια, τα ανατολικά και τα δυτικά της Ευρώπης ε, Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια επικοδομητική έκθεση που να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές, ε, λαμβάνοντας υπόψη την αστική εξάπλωση για παράδειγμα που δυσκολεύει τη δημιουργία ενός ε, δικτύου ε, ενταξιακού, αποτελεσματικού και ασφαλούς. Νομίζω ότι έτσι έχω συνοψίσει τα περισσότερα θέματα. Ξέρω όμως ότι κάποιοι συνάδελφοι θα θέλουν να αναπτύξουν κάποια από αυτά τα σημεία περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τσοζονόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια που μας παρουσίασε αυτή την έκθεση. ως πρώην δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης της τσεχικής ε, ε, δημοκρατίας και ως κυβερνήτης μιας περιφέρειας ε, ασχολήθηκα για 16 χρόνια με την αστική κινητικότητα και έχω την εντύπωση ότι πρέπει εδώ να είμαστε ρεαλιστές διότι Κάποια στοιχεία είναι υπερβολικά ε, στραμμένα προς το μέλλον και δεν ξέρουμε τι θα γίνει εντωμεταξύ με τις νέες τεχνολογίες ε, κτλ. Είναι δύσκολο κανείς να μαντέψει τι θα γίνει στο μέλλον. Πιστεύω πως κάθε αστική πόλη έχει ιδιαιτερότητες διαφόρων ειδών. Δεν υπάρχουν δηλαδή λύσεις ε, που να ταιριάζουν σε όλες τις πόλεις. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε έκκληση στην επικουρικότητα. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο για όλες τις πόλεις, όπως αποδεικνύεται από τη δική μου τουλάχιστον εμπειρία στη διάρκεια όλων αυτών των ε, ετών. Ε, αν προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η ιεραρχία των διαφόρων ε, ειδών ε, μεταφορών, όπως προσπάθησε να το κάνει και η συγχύτρια. Ε, θα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γιατί δεν έχει παντού νόημα να έχουμε ας πούμε πεζοδρόμους ή ποδηλατόδρομους γιατί σε ορισμένες ε, περιοχές αυτό δεν ε, γίνεται, ενώ έχουν ε, αλλού γίνει προσπάθειες για ποδηλατόδρομους ε, ή για ποδηλατόδρομους, αλλά δεν έχει όμως λειτουργήσει πάντοτε αυτό το πρόγραμμα. Όταν μιλάμε για ουδετερότητα κλιματική, έχω την εντύπωση ότι ευνοούμε τον ηλεκτρισμό ως ε, πηγή ενέργεια. Δεν ξέρω όμως αν αυτό έχει κάποιο νόημα πραγματικό, γιατί και ο ηλεκτρισμός έχει παρενέργειες. Πρέπει να ενισχυθούν τα δίκτυα ηλεκτρισμού και κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά περίπλοκο στις πόλεις. Και μέσα στις μεγάλες πόλεις πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να ενισχυθούν τα ε, δίκτυα. Άλλες τώρα εναλλακτικέ. που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να στηριχθούν αυτές οι τεχνολογίες που δεν έχουν ε, επιβαρυντική θετικό αποτέλεσμα στο περιβάλλον. Επίσης, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ε, αστική κινητικότητα, αλλά χωρίς αυτό να προδιαθέτει την κατανομή κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιστήσω την προσοχή σας ότι όταν χρησιμοποιούμε τέτοια κονδύλια Είμαι σύμφωνος, αλλά δεν θα πρέπει να βάζουμε υπερβολικά πολλά χρήματα ε, στην άκρη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για τις τροπολογίες βεβαίω θα σας υποβάλλω. Χαίρομαι για τη συνεργασία και με χαρά, τα χαρά θα συμμετέχω ε, στις ε, συναντήσεις με τους και ηγητές και στη μελλοντική συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ja, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά που είναι η γλώσσα των πολλών ποδηλατών που πάνε στην Ολλανδία στη δουλειά τους με το ποδήλατο. Όταν μιλάμε για αποτελεσματική και βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις, δεν συμφωνούμε για το τι είναι, αλλά δεν συμφωνούμε για το πώς θα το καταφέρουμε. Συχνά τα ακούμε αυτά, συχνά ακούμε το θέμα της επικουρικότητας. Η εισηγήτρια σίγουρα δεν έχει εύκολη δουλειά να κάνει. Σχηνοβατή Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ε, τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι αυτός θα πρέπει να είναι ένα σε, ε, γνώμονας δεν θα πρέπει να είναι ένας όρος τον οποίο εμείς επιβάλλουμε και αποφασίζουμε γιατί υπάρχουν διάφορα επίπεδα στην Ευρώπη υπάρχουν ε, οι πόλεις ε, οι επαρχίες, υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα και πρότυπα και σίγουρα υπάρχουν κάποιες ε, πόλεις που αποφασίζουν για τις ε, πόλεις αλλά για τις ίδιες τις συνθήκες αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβάλλουμε ένα σχέδιο για την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Οι αρμοδιότητες ε, για αυτά τα θέματα ε, τοποθετούνται σε διαφορετικό επίπεδο σε κράτος μέλος και αυτό ε, σημαίνει τη διαφορά. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι το να ενταχθεί η αστική κινητικότητα στο ΣΕΦ και στο ΤΕΝΤΗ. Ναι, πρόκειται Ε, δεν θα πρέπει να δούμε ακόμα περισσότερα κατόφλια, ακόμα περισσότερα σχέδια από την ε, ΣΕΦ που ήδη έχει εγκριθεί. Εγώ θα ήθελα να παραμείνω τα πράγματα ως έχουν για τα διαρθωτικά προγράμματα, γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθούν ε, δυσκολίες. Έπειτα, σε μια έκθεση του Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να μιλάμε για απαγορεύσει ή για αποκλήσει ή για εξαιρώσει. Ίσως πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να μην ε, δώσουμε μια συγκεκριμένη ιεραρχία των τρόπων μεταφορών ε, να μην επιβάλλουμε κάτι για τις δημόσιες μεταφορές ή για την ανώτατη ταχύτητα, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία αποφασίζονται ανάλογα με την πόλη. Ας πούμε, δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλους. Είναι μία ε, λύση κάθε φορά συγκεκριμένη ε, που Ισχύει χωριστά για την κάθε πόλη. Οι όσοι θέλουν να χρησιμοποιούν τις, τα μέσα μαζικής ε, ε, μαζικών μεταφορών θα πρέπει αυτή να αποφασίζουν. Ας πούμε στην Ολλανδία ασκήθηκε ειδική πολιτική με, τις, ε, με τα ποδήλατα, με συνδέσεις, ε, συνδέσεις με τα δίκτυα που λειτουργούν στην εντέλεια. Για παράδειγμα, στα φανάρια υπάρχει χώρος προτεραιότητας για τα ποδήλατα ας πούμε, σε σχέση με τα λεωφορεία. Εμείς το αποφασίσαμε έτσι. Ε, δεν μπορούμε να υποβάλουμε όμως την ίδια ιεραρχία σε όλους. Ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε έξυπνες λύσεις για την αστική κινητικότητα. Τώρα, ITS, ΦΥΗ, ε, e, συστήματα μεταφορών. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι θα πρέπει αυτά να εντάσσονται στις ΦΥΗς πόλεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν λύσεις ευφυών μεταφορών, χρειάζονται χρήματα, λεφτά από τα κοινοτικά ταμεία, αλλά με ανησυχεί κάπως και ο ορίζοντας 2020, το οποίο στην ουσία ε, ε, ε από το πρόγραμμα Juncker. Ας πούμε προγράμματα που είχαν στόχο την έρευνα, Όσον αφορά δηλαδή τα οχήματα που, επικοινωνούν μεταξύ τους και που επικοινωνούν με το περιβάλλον γύρω τους όσον αφορά τις, επιδο... επιδοτήσεις ε, ε, ή το σχέδιο για ηλεκτρική φόρτιση, όλα αυτά με ανησυχούν που δεν μπορούμε να τα κάνουμε τώρα. Πρέπει οπωσδήποτε να τα συζητήσουμε γιατί κατά τη γνώμη μου το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και ευφυείς λύσεις αφορούν τους χρήστες των μεταφορών στις πόλεις και καθορίζουν το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Κοίταξια ρεπορτέρη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Ντελή, την εισηγήτρια να είμαστε προσεκτικοί για το θέμα αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Μεταφορών. Και λέω να είμαστε προσεκτικοί γιατί πρέπει να ε, καταφέρουμε να βρούμε τις σωστές λύσεις, να καταλήξουμε στη σωστή έκθεση. Να μην έχουμε μόνο περιορισμούς και απαγορεύσεις, να, αλλά να προσφέρουμε εναλλακτικέ. Να προσπαθήσουμε να ε, αναπτύξουμε έναν σχεδιασμό των ε, ρυθμίσεων των μεταφορών, των εισιτηρίων, των τρόπων έκδοσης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες μορφές μεταφορών. Στόχος μας πρέπει να είναι να δώσουμε κίνητρα, ε, να ενθάρρυνση για χρήση των μέσων μεταφοράς που εμείς θέλουμε. Το πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε το κλίμα, τις ε, εναέριες μεταφορές. Είναι κάτι το καθαριστικό. Να βρούμε τη σωστή ισορροπία για να ε, υπάρξει στήριξη στην έκθεσή μας να στηρίξουμε την ανάπτυξη του μεταφορικού σχεδιασμού στις πόλεις σε όλη την Ευρώπη και να διασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των επίπεδων διακυβέρνησης, τοπική, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και εθνικό κεντρικό κράτος. Να βρούμε σωστό σημείο ισορροπίας, να βρούμε τις λύσεις με κίνητρα, όχι με αντικίνητρα, με θετικά μέτρα, με καταφατική δράση. Έτσι θα λειτουργήσουμε ε, πολύ πιο γρήγορα από το να ρυθμίζουμε κανονιστικά τα πράγματα και να τα απαγορεύουμε από το νόμο. Από εκεί και πέρα. Πώς θα το οργανώσουμε αυτό σε όλη την Ευρώπη. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος δεν θα θέλει να μπει στο δικό του αυτοκίνητο, ότι ο κόσμος θα ξέρει και θα βλέπει ότι έχει εναλλακτικέ. Πώς θα τους μειώσουμε την ανάγκη να μετακινηθούν δια του ιδιωτικού αυτοκινήτου από το ένα μέρος στο άλλο. Ε, πρέπει να μπορούμε να έχουμε υπόψη μας ότι στα διαφορετικά κράτη-μέλη, στις τόσο διαφορετικές περιφέρειες και, και πόλεις, πρέπει ο καθένας να βρει το δικό του τρόπο να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω λοιπόν ότι με τους σκιώδεις εισηγητές θα εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα και θα τα αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προέρχομαι από μια χώρα αρεοκατοικημένη, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τις υπαίθριες μεταφορές. Ακούστηκε ότι θα είναι πολύ ωραίο να έχουμε σιδηρόδρομους ε, για να κάνουμε τα ψώνια μας, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν. 50 ε, τόνους ε, προϊόντα την ημέρα μπορεί να λαμβάνει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ε, αυτό όμω δεν μπορεί να γίνει με ποδήλατο. Ε, πώς μπορεί κανεί να μεταφέρει κατεψυγμένα με ποδήλατο ή με λεωφορείο. Ε, βλέπω εδώ μία αφέλεια σχετικά με το πώς λειτουργούν οι μεταφορές στο τομέα της εφοδιαστικής. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο περιβάλλον, θα πρέπει όμως από την άλλη να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα θα πρέπει να είναι σημαντικές οι φιλοδοξίες μας, ε, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και την πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε έρευνες για εναλλακτικά καύσιμα. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μεταφορές χωρίς να επιβαρύνουμε επιπλέον ε, το ήδη επιβαρημένο περιβάλλον μας. και ένας τρόπος ε, να λύσουμε κάποια προβλήματα είναι οι μεταφορές εμπορευμάτων ε, να γίνονται τη νύχτα. Στην ε, Δανία, με, στη Σουηδία, συγγνώμη, με 20 πόντους χιόνι και θερμοκρασία μείων 10 βαθμούς είναι αρκετά τα προβλήματα. Μα ενδιαφέρουν λοιπόν οι ποδηλάτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να επενδύσουμε ε, στα καλύτερα καύσιμα. Σήμερα έχουμε για παράδειγμα λεωφορεία με ντίζελ και βέβαια έχουμε ε, μεταφορές ε, όπως οι άλλες χώρες το καλοκαίρι, αλλά τον χειμώνα είναι άλλες οι κλιματικές συνθήκες τα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά για τα βαρέα οχήματα είναι δύσκολο να έχει κανείς ε, επαρκή χωρητικότητα στις ε, μπαταρίες. Νομίζω όμως ότι θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να έχουμε μικρά φορτηγά ηλεκτροκίνητα. και βέβαια είναι πολύ ωραία τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, αλλά χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι λοιπόν σημαντικό και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο να γίνεται με τρόπο φιλικό προ το περιβάλλον. Δεν, δεν έχει νόημα να έχουμε καθαρέ πόλει, εάν έχουμε πολλή ρήπανση εκεί που παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίσω το χρόνο ομιλία σε δύο λεπτά. Κλάουδια Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω γρήγορα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την έκθεση. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν σημαντικά θέματα όπως είναι η κλιματική στόχη, οι στόχοι της Λευκής Βίβλου κλπ. Θέλουμε βιώσιμε λύσεις και θα μπορούσα να δεχθώ να έχουμε ευρωπαϊκούς ποδηλατόδρομους. Ε, προέρχομαι από μια πόλη της Αυστρίας η οποία είναι η πιο φιλική προς το ποδήλατο εντός της Αυστρίας, το Σάλτσπουργκ. Έχουμε πολλούς ποδηλατόδρομους, έχουμε ζώνες ε, συνάντησης, έχουμε ζώνες ε, για τους πεζούς έχουμε και η ηλεκτροκινητικότητα σε συνεργασία με ε, διάφορες εταιρείες και ε, θα πρέπει να επικρίνω όταν η έκθεση γράφει ότι η πόλεις ε, με πολλούς πεδηλατόδρομους, ε, δεν έχουν τόσο καλή κινητικότητα. Δεν μ' αρέσει που η έκθεση έχει ύφος διδακτικό και θεωρεί ότι μόνο με έναν τρόπο μπορεί να έχουμε βιώσιμη κινητικότητα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας καλέσω να λάβουμε υπόψη και τις πόλεις, διότι ε, αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τις πόλεις ε, θα αποτύχουμε. Οι πόλεις θα μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και δεν νομίζω ότι είναι δουλειά της Κομισιόν να εκπονεί οδηγίες σχετικά με διάφορες λεπτομέρειες. Να μην έχουμε λοιπόν ύφο διδακτικό για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, πέρα Τερμόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους σκιώδης εισηγητές για τη θετική αυτή δουλειά που έκαναν, αλλά και για τους στόχους που έχουν ορίσει, την προσοχή για το περιβάλλον, την προσοχή ε, για τα κοινωνικά ζητήματα. Ίσως θα πρέπει να απομακρυνθούμε λίγο από την αντικειμενική προσέγγιση ε, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια πιο καθολική προσέγγιση. Και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τα αυτοκίνητα, αλλά να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καινοτόμα διαχείριση της αστικής ε, κινητικότητας ε, ας πούμε, αν σκεφτεί κανείς πόσους γύρους κάνει κανείς για να βρει θέση πάρκινγκ. Ε, θα πρέπει να μειωθεί 10 με 18% η μείωση των, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τα αίτια που είναι η συγκέντρωση των μέσων, ε, η ταχύτητα, η ποιότητα των συστημάτων ασφάλειας, το θέμα των υποδομών, το σύστημα των στάσεων και των πάρκινγκ. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα του της... Ε, γιατί αν σκεφτούμε τον δίζελ νέας γενιάς έχουμε εκπομπές που είναι παρόμοιες με αυτές του μεθανίου. Και άλλη μια σκέψη είναι αυτή <coughs> που συμπίπτει με μια καθολική προσέγγιση, δηλαδή την άπεψη του σχεδιασμού, του αστικού σχεδιασμού, της πολεοδομίας και του συνδυασμού αυτής με τις μεταφορές. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα της ε, ευφυΐες, Υπάρχουν ευφυΐ προγράμματα όπως ας πούμε το Φράιμπουργκ που είναι μια οικολογική πόλη και εγώ πιστεύω ότι εφόσον θέλουμε να μιλήσουμε για πρότυπα είναι ένα από αυτά και να πούμε ας πούμε για χάρτες επάρκειας ε, των πόλεων, ε, εγχειρίδια των ευφυών πόλεων και αυτό που έχουμε και στην Ιταλία, το, ε, τις εικονικές αυτές και ενάρετες λύσεις που συνδυάζουν τις πόλεις με τις υφείς μεταφορές. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, διότι η έκθεση περιέχει πολύ σημαντικά στοιχεία. Προστασία του περιβάλλοντος, μείωση των εκπομπών. Και εκτιμώ ε, την αδιαλαξία σας, αλλά δεν συμφωνώ με κάποιες από τις συμβαστικές προτάσεις όσον αφορά τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς. Πιστεύω ότι η ισορροπία σημαίνει να υπερασπίζεται κανείς τη θέση του, αλλά να σέβεται και τις απόψεις άλλων. Σημαντικό λοιπόν είναι να παραμείνουμε λογικοί, να λάβουμε υπόψη μας τις δυνατότητές μας και να λάβουμε υπόψη μας και την πολυπλοκότητα του θέματος. Οι πόλεις εντός της Ευρώπης διαφέρουν πολύ η μία από την άλλη. Θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον, ε, την επόμενη 15 ετία ή 20 ετία. Θα πρέπει όμως όλα αυτά να αποτελέσουν μια διαδικασία θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει τι συνέπειες έχει η μόλυνση του περιβάλλοντος, πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία των ανθρώπων με αντικειμενικές έρευνες. Θα πρέπει και οι δήμαρχοι των πόλεων να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, διότι αν δεν συμμετάσχουν ε, με όλη την καλή μας βούληση δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Πριν κάποιες εβδομάδες ακούσαμε ότι υπήρχε οξία ατμοσφαιρική ρήπανση στο Λονδίνο και ο Δήμαρχος είπε μην ε, πάρετε το αυτοκίνητο για κάποιες μέρες. Ε, δεν υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Λονδίνο, αφορά και άλλες μεγάλες πόλεις. Ελπίζω η έκθεση αυτή τελικά να αποτελέσει καλό συμβιβασμό ε, και να έχουμε καλά αποτελέσματα για τους πολίτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Ντίτερ Κόχ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, κύριε Αντελή, να σας ευχαριστήσω για την έκθεση σας. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά λόγω του περιορισμού του χρόνου θα ήθελα να αναφέρω τρεις πτυχές που θα ήθελα να δω στην έκθεσή σας. Καταρχάς ε, το, το ticketing στην πολυτροπικότητα. Δεύτερον, ε, τα ευφυή e e συστήματα μεταφορών και την ε, διαβίου εκμάθηση των πολιτών μας, ε, διότι εάν δεν μάθουν να χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά, τότε δεν ε, θα πετύχουμε τίποτα. Και τρίτον, είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα του τουρισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κριστίνη Ριβονταλό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Καρήμα, του σκιώδεις εισηγητές και κυρίως την κυρία Άντερσον για την παρουσίαση και την οπτική γωνία που έχει οθετήσει αυτή η εξαιρετικά σημαντική έκθεση. Συμφωνώ απολύτω με του προλαλήσαντε. Να επιμείνω όμω σε ένα σημείο που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη βελτίωση τη προσβασιμότητα. Η έννοια της βιωσιμότητας να ιδωθεί και υπό την κοινωνική οπτική γωνία. Δεν έχουμε μόνο την περιβαλλοντική διάσταση και τον κίνδυνο δημόσιας υγείας. Έχουμε και την πρόκληση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Θα πρέπει η δημόσια υπηρεσία μεταφοράς να αναδειχθεί, να αναβαθμιστεί για να έχουμε περισσότερη κοινωνική συνοχή. Συμφωνώ με την Καρίμα και τη Λούση. Πρέπει να προωθήσουμε τις προκτήσεις της αστικής κινητικότητας σε συνέργεια με την COP21, την προπαρασκευαστική διάσκεψη για το κλίμα ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και καλώ τις υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πούν σε ποια κατάσταση, σε ποιο σημείο είναι οι πρωτοβουλίες σας Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα Σχέδια Αστικής Κινητικότητας. Όλα αυτά εντάσσονται στο πακέτο για την αστική κινητικότητα που εγκρίθηκε το 2013. Πώς αξιολογεί η Κομισιόν την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την Καινοτομία, έξυπνες πόλεις και κοινότητες για ε, τις υποχρεώσεις της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης αυτή η εταιρική σχέση να είναι πιο ορατή και να εφαρμοστεί στην πράξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που τηρήσατε και τον χρόνο. Ζήτησα το λόγο, διότι αν δεν λάβουμε υπόψη μας σε την αστική κινητικότητα, δεν πρόκειται να σταματήσουμε την αλλαγή του κλίματος. Θέλουμε κινητικότητα, θέλουμε όμως να προστατεύσουμε και το κλίμα. Πώς ε, θα γίνει αυτό. Κανείς ε, δεν θέλει να απαγορεύσει τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να βρούμε άλλη πολιτική μεταφορών και πώς θα την εφαρμόσουμε. Δεν χρειάζεται να περιορίσουμε την κινητικότητα. Τα τελευταία 100 χρόνια βλέπουμε ότι τίποτα δεν ε, έχει αλλάξει στην κινητικότητα, διότι δύο ή τρεις φορές τη μέρα ο κόσμος εγκαταλείπει το σπίτι του. Μόνο οι αποστάσεις έχουν γίνει μεγαλύτερες, όχι όμως η κινητικότητα αυτή καθ' αυτή. Αυτό το δείχνει μια έρευνα. Επίσης, έχουμε τεράστιες δυνατότητες στην, ε, στο Βερολίνο. Ε, υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι με ποδήλατα ε, φορτηγά μπορούν να καλύψουμε μεγάλο μέρος των μεταφορών εμπορευμάτων. Οι επενδύσεις δεν είναι μόνο λίγες. Έχουμε το χάσμα των επενδύσεων, ε, έχουμε όμως και λάθος επενδύσεις. Στο Βερολίνο βλέπουμε ότι ε, σε 30 χρόνια χτίστηκαν 3 ε, χιλιόμετρα μετρό, ενώ με τα ίδια λεφτά θα μπορούσαμε να έχουμε 120 χιλιόμετρα δρόμων. Αυτή δεν ήταν η καλή απόφαση κατά τη γνώμη μου. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, η χρήση της γης είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πώς μπορούμε να κάνουμε σωστό σχεδιασμό. Θα πρέπει κάποιες ε, χώρες να τις ε, σχεδιάσουμε διαφορετικά. Μπορούμε να συγκρίνουμε την Ατλάντα με την Βαρκελόνη που έχουν τον ίδιο αριθμό πολιτών. Επίσης, όσον αφορά την επικουρικότητα, αν ε, οι πόλεις δεν λαμβάνουν ευρωπαϊκό χρήμα, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν μπορούμε ως Ευρώπη να τους δίνουμε τα χρήματα ε, και να τα χρησιμοποιούν για ανόητα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε τι γίνεται με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Τελευταία παρατήρηση. Κύριε Τολνόφσκι, σας παρακαλώ ακούστε με. Αναφερθήκατε στους ποδηλατόδρομους. Ε, στο Βερολίνο πριν από 25 χρόνια, το 80 ε, των δρόμων έγινε μικτός, έγιναν μεικτοί δρόμοι για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Κανένα ε, δεν το αφισβήτησε αυτό, αλλά θα πρέπει κανείς να εξετάσει την κατάσταση. Και Πίτερ Λούπκι, ε, ε, στο Όσλο είδα ποδηλάτες που και το χειμώνα μου είπαν ότι παίρνουν το ποδήλατο. Γίνεται λοιπόν η κυρία Κοπτσίνσκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό απόγευμα κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση που μόλις ακούσαμε αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το θέμα των πόλεων και το θέμα της αστικής κινητικότητας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ. Και όπως λέει η συγγήτρια στην έκθεσή της, την οποία εκτιμούμε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αστική κινητικότητα λόγω των σημαντικών στόχων της απαλλαγής της οικονομίας από εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και βελτίωση της ποιότητας. Θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε με την αστική κινητικότητα, διότι και οι μεταφορές ε, αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των πόλεων. Στις πόλεις μένουν οι περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις πόλεις παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Θα πρέπει να εξετάσουμε αναλυτικά το θέμα αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά που είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να, να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επί πολλά χρόνια στηρίζει τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση της αστικής κινητικότητας στην Ευρώπη από την εισηγήτρια αλλά και από αρκετούς ευρωβουλευτές της Επιτροπής άκουσα σήμερα ότι υπάρχει ανάγκη να αναλυφθεί δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Θα πρέπει να είναι σαφής η θέση μας Υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσουν οι πόλεις το θέμα της αστικής κινητικότητας. Είναι όμως πολύ σημαντικό θέμα και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε στην τύχη τους της πόλεις. Υπάρχουν ε, διάφορες δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Κάποιες είναι καθήκοντα των δημάρχων, άλλες είναι των περιφερειακών και εθνικών.